Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Προσέξτε παρακαλώ, πρόσχομεν. Σας καλωσορίζω σε αυτή την ακρόαση για την ισότητα των φίλων. Λέγομαι Αντιγόνη Παπαδοπούλου και προεδρεύω εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης, της οποίας είμαι και μέλος. Δυστυχώς η κυρία Περβάνς δεν θα προσέλθει διότι είχε ανηλυμένη υποχρέωση και αυτό την αντικαθιστώ. Αριστερά μου είναι η Ρετζίνα Μπάστος που αντιπροσωπεύει την Επιτροπή των Γυναικών. Θα συμπροεδρεύσομεν λοιπόν. Επιτρέψτε μου καταρχήν να σας πω μερικά λόγια έτσι εισαγωγικά για την ακρόαση αυτή. Work-life balance and gender equality. Πιστεύουμε ότι αυτή η εξισορρόπηση πετυχαίνει πολλούς από τους ενωσιακούς στόχους όπως την απασχόληση και την ισότητα στην απασχόληση ανδρών και γυναικών, προωθεί την ανάπτυξη των παιδών και φυσικά ενθαρρύνει και την ισότητα των φύλων. Η εξισορρόπηση αυτή της ε, κοινωνικής δουλειάς ή της εμπειρίας εργασίας είναι κάτι που διευκολύνει και τους γονείς και την ανατροφή των παιδών. Η ελαστικότητα, η μερική εργασία, ελαστικές συνθήκες εργασίας επίσης μπορούν να διευκολύνουν τα πράγματα. Θέλουμε να καθοριστούν κανόνες για την προώθηση των βελτίστων πρακτικών που να βελτιώνουν την κατάσταση αυτής της ενίας work-life balance. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι το πρώτος γύρος των συζητήσεων που λέγεται work-life balance ως παράγον της ισότητας των φύλων θα σε αυτήν θα προεδρεύει η κυρία Μπάστος και θα μιλήσουν η κυρία Κλάουδια Μένε που είναι συνομοσπονδιακή γραμματεύς της Ευρωπαϊκής ΓΕΣΕ, κυρία Κωνσταντίνα Νταβάκη που είναι ερευνήτρια από το London School of Economics και επίσης η κυρία Άκνες Παρενφίλιον προγραμματίστρια για τις συνθήκες εργασίας στο Eurofound. Στο τέλος των παρουσιάσεων θα γίνει μία σειρά ερωταπαντήσεων και μετά θα οργανωθεί ο δεύτερος γύρος που θα λέγεται η εργασία και οικογενειακή ζωή. Θα μιλήσουν η κυρία Γόλμιν Μπέντλερ, πρόεδρος του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου και η κυρία Άννα Ρούπιν από το Σουηδικό Αριστερό Κόμμα. Και βέβαια και εκεί θα υπάρξουν ερωταπαντήσεις. Και ύστερα τα συμπεράσματα, η κυρία Ρετζίνα Μπάστονς και τα τελικά συμπεράσματα εγώ. Αυτό είναι το πρόγραμμα και τώρα θα δώσω το λόγο αμέσως στη συνάδελφο από την Πορτογαλία Ρεγκίνα Μπάστος που εκπροσωπεί και την Επιτροπή Γυναικών. Ευχαριστώ. Πρόεδρε και συνάδελφοι κύριε Παπαδοπούλου, είμαι η Ζωζίνα Μπάστου, εκπροσωπώντας την πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών, κύριο Γκούσταυσον, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ε, συνεδρίαση στον ΟΗΕ για την κατάσταση των γυναικών. Σας καλωσορίζω όλους. Το θέμα της ακρόασης είναι πώς θα συνδιαλέξουμε την οικογενειακή με την εργασιακή ζωή. Ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό για την ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή μας. Κατά τη διάρκεια της θητείας μας προσπαθήσαμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία του θέματος αυτού και να προωθήσουμε την καλύτερη δυνατή πρακτική ούτως ώστε να υπάρξει όσο καλύτερη ισορροπία γίνεται μεταξύ των δύο αυτών ε, διαστάσεων, δουλειά, οικογένεια και δουλειά, πάντα σε ένα πλαίσιο σεβασμού της ισότητας των φύλων. Το 2009 και μετά το Κοινοβούλιο υπέβαλε μια σειρά εκθέσεων για το θέμα αυτό και ένα ψήφισμα για την ισότητα ευκαιριών. Μια δεύτερη νομοθετική δραστηριότητα αφορούσε τις γυναίκες στον τομέα των υπηρεσιών. Ένα ψήφισμα για την κατάργηση των στερεότυπων ε, βάση φύλου στην Ένωση. Στην Ένωση, συγγνώμη. Πολλοί αυτή τη στιγμή στην Ένωση υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι που δεν είναι ικανοποιημένοι από το πώς μπορούν να συνδυάσουν οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Οι γυναίκες περισσότερο από όλου, γιατί έχουν περισσότερες οικογενειακές ευθύνες σε σχέση με τους άνδρες γενικά. Πολύ συχνά οι γυναίκες ασχολούμενοι με τα παιδιά και την ανατροφή τους δίνουν λιγότερο χρόνο στην επαγγελματική τους δραστηριότητα, κάνουν μερική απασχόληση με μικρότερη ασφάλεια στο, στη σταδιοδρομία, στη τους και λιγότερες παροχές. Οι άνδρες δουλεύουν περισσότερο, ακόμα και όταν έχουν μικρά παιδιά, δίνοντας λιγότερο χρόνο στην οικογένειά τους. Η ισορροπία λοιπόν μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακή ζωής είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, κομβικό για την Επιτροπή Γυναικών, αλλά και για την Επιτροπή απασχόληση ταυτόχρονα. Στην πρώτη αυτή στρογγυλή τράπεζα της ακρόασης θα ασχοληθούμε με την ακρόαση για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Έχουμε τρεις εμπειρογνώμονες μαζί μας. Να ευχαριστήσω και τις τρεις εμπειρογνώμονες και να θυμίσω ότι κάθε μία από αυτές έχει ένα δεκάλεπτο που θα παρακαλούσα να σεβαστούν. Μετά θα γίνει μια συζήτηση. Δίνω αμέσως το λόγο στους διάφορους εμπειρογνώμονες. Αφού μίλησε η κυρία Παπαδοπούλου πρώτα. Η Κλαούδια Μένε τώρα έχει το λόγο, είναι ομοσπονδιακή γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνδικάτων. Ξέρουμε ότι θα φύγει, θέλει να φύγει στις τέσσερις και χαρά την έχουμε μαζί μας για να μοιραστούμε μαζί της τις εμπειρίες της. Είχαμε καλέσει την κυρία Μένε σε πολλές περιπτώσεις και σε ένα εργαστήρι που είχαμε διοργανώσει όταν γινόταν λόγος ακριβώς για το πώς ε, θα μπορούσαμε να εξορροπήσουμε καλύτερα την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή και το 12 όταν συζητούσαμε για τη συμμετοχή γυναικών στην αγορά εργασία. Κατόπιν εξελέγει το, 2000, το Μάιο του 2011 Γενική Γραμματέας ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Συνδικάτων με θέμα ακριβώς την ισότητα των φύλων. Ασχολείται με τις δημογραφικές αλλαγές ιδιαίτερα. Την ευχαριστώ που είναι εδώ μαζί της και της δίνω το λόγο. thank you, Mr. Chair, and all the other... Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ευρωβουλευτές ε, και κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ε, καλωσορίσω και την Επιτροπή Γυναικών ε, της Ευρωπαϊκής ε, Ομοσπονδίας Μεταφορών, διότι και εγώ είμαι εργαζόμενη στον τομέα αυτόν. Ε, ανήκω βέβαια στην Ένωση της Γερμανίας. Με κάλεσαν εδώ να μιλήσω για την ισορροπία επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου και Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο πλαίσιο και να σας πω γιατί θεωρούμε σημαντικό να εξετάσουμε τις πολιτικές αυτές, ακόμα και αν ε, θεωρήσετε ότι οι πολιτικές ε, συμφιλίωσης ε, ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου είναι μια παλιά συζήτηση επειδή έχουμε πολλές πολιτικές τώρα πια έχουν εφαρμοστεί μέτρα. Παρ' όλα αυτά παραμένει ψηλά στο θεματολόγιο μας και θα σας πω γιατί πιστεύω ότι ε, Επίγει να εξετάσουμε το θέμα αυτό. Βρισκόμαστε σε μια κρίση. Η κρίση, κατά τη γνώμη μας, δεν έχει περάσει και ιδιαίτερα οι συνέπειες ε, για την κοινωνία και την ε, αγορά εργασίας είναι ανησυχητικές. Γι' αυτό σήμερα γίνεται μια διάσκεψη κορυφής συνδικαλιστικών οργανώσεων που πραγματοποιείται σήμερα και θα πρέπει να παρευρεθώ εκεί αργότερα. Έχουμε λοιπόν υψηλή ανεργία, υψηλό ποσοστό φτώχειας και τα στοιχεία του Φεβρουαρίου δείχνουν ότι πάνω από το 30% του πληθυσμού ε, σε ηλικία εργασίας ε, ε, θεωρείται ότι βρίσκεται κάτω από το όριο της και ιδιαίτερα οι γυναίκες. Ε, πέφτουν τα ποσοστά γεννήσεων και οι ε, πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί σημαίνουν ε, ότι έχουμε μακρύτερη επαγγελματική σταδιοδρομία σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Ο κόσμος πρέπει να εργάζεται μέχρι τα 72 του χρόνια. Γιατί λοιπόν αυτό είναι θέμα των δύο φύλων και θέμα που σχετίζεται με τη μειονεκτική θέση των γυναικών. Έχει αναφερθεί ότι οι γυναίκες ε, εργάζονται σε μεγάλο βαθμό με μερική απασχόληση και αν ε, εξετάσετε την κατάσταση των οικοκυριών ε, θα διαπιστώσετε ότι οι γυναίκες που ζουν, που συμβιώνουν, θεωρούνται πιο προστατευμένες από ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες, επειδή έχουν και κάποιο άλλο εισόδημα, αλλά βρίσκουμε ότι έχει διαβρωθεί το πρότυπο αυτό, διότι και οι άντρε βρίσκονται επαγγελματικά σε όλο και πιο επισφαλή θέση και αν κοιτάξετε τα στατιστικά στοιχεία της κρίσης θα διαπιστώσετε ότι Ε, ότι τα ποσοστά δείχνουν ε, ότι τα κενά φαίνεται να ε, κλείνουν, αλλά αυτό δεν οφείλεται σε καλύτερες συνθήκες ε, του αντίον ε, αντιπροσωπεύουν εξίσωση προς τα κάτω. Δηλαδή και οι άντρες αντιμετωπίζουν όλο και πιο επισφαλείς θέσεις εργασίες σε μείωση των μισθών τους κλπ. Αυτή λοιπόν η κατάσταση είναι ανησυχητική για μας. Τι βλέπουμε λοιπόν ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποφάσισα να σας παρουσιάσω όχι μόνο μια επισκόπηση του πώς το βλέπουμε εμείς ως συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ε, σας ε, παραπέμπω εδώ σε στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου του 2013. Δεν είναι πολύ εύκολο να τα διαβάσετε, αλλά θεώρησα ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ε, να κοιτάξουμε αυτό το Ευρωβαρόμετρο, διότι τα στοιχεία αυτά ε, συλλέχθηκαν στο πλαίσιο μιας έκθεσης ε, που ε, κοπώνησε το Κοινοβούλιο σχετικά με τις συνέπειες της κρίσης. Βλέπετε εδώ λοιπόν ότι οι γυναίκες, πώς βλέπουν οι γυναίκες και άντρες την κατάσταση. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι πολιτικές συμφιλίες επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου καθώς και η ψαλίδα στις αμοιβέ είναι προβλήματα που έχουν επιδεινωθεί με την κρίση. Από τη μία λοιπόν έχουμε στατιστικά στοιχεία ότι φαίνεται να γινόμαστε πιο ίσοι, αλλά οι πολίτες θα σας πούν ότι η πραγματική εικόνα είναι διαφορετική, ε, έχουμε ε, σημαντικά προβλήματα. Δεν είναι εύκολο να διαβάσετε τα στοιχεία στην οθόνη. Αλλά η τελευταία διαφάνεια που ήθελα να σας δείξω δείχνει ότι οι νέες γυναίκες, ε, το περισσότερο από το 50 60% των ε, νέων γυναικών σε 17 έως 35 ετών ε, θεωρούν ότι το σημαντικότερο πρόβλημα για αυτές είναι ότι οι εργοδότες κυρίως κοιτάνε αν έχουν παιδιά ή όχι. Ενώ στους άντρες εξετάζουν περισσότερο τις δεξιότητες και τα προσόντα τους. Το πρώτο κριτήριο λοιπόν για την πρόσληψη γυναικών είναι η οικογενειακή τους κατάσταση. Απομένουν λοιπόν πολλά να γίνουν, ιδιαίτερα όσον ε, αφορά την, τον συνδυασμό ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου, κυρίως όταν μιλάμε για οικογένειες με παιδιά. Αποτελεί μια μακροπρόθεσμη δέσμευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις όμως σε όλα τα επίπεδα, περιφερειακό, τομεακό, τοπικό, εθνικό, ασχολούνται με το θέμα αυτό. Δεν μπορώ να σας δώσω τον πλήρη κατάλογο, αλλά θα ήθελα να αναφέρω ότι εμείς η ΕΤΥΚ μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο εργαζόμαστε συνεχώς πάνω στο θέμα αυτό. Ένα από τα βασικά επιτεύγματά μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η γηγονεακή άδεια που βασίζεται σε μια συμφωνία των κοινωνικών εταίρων του 1996 που αναθεωρήθηκε το 2010. Ε, ακόμα βρισκόμαστε στη διαδικασία επικύρωσης. Κάποια κρατημέλη μόλις πέρσι επικύρωσαν ε, τη σχετική οδηγία. Έχουμε μια αυτόνομη ε, συμφωνία για την εργασία εξ και έχουμε μια άλλη για την ε, μερική απασχόληση, όπου εξετάζουμε το θέμα του συνδυασμού οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Άλλος σημαντικός τομέας για μας είναι η πολιτική για την ε, ισότητα των δύο φύλων. Έχουμε τέσσερις προτεραιότητες. Ε, μία από τις προτεραιότητες εδώ ήταν ακριβώς ε, ο συνδυασμός ιδιωτικού και, και επαγγελματικού βίου και θα γίνει μια διάσκεψη φέτος τον Ιούνιο. Εξετάζουμε εδώ τις τις λύσεις που μπορούν να παρασχεθούν σε επίπεδο επιχείρησης οι περισσότερε δραστηριότητε που πραγματοποιούνται σε επίπεδο ε, επιχειρήσεων έχουν να κάνουν ακριβώ με τέτοιε πολιτικέ για να διευκολυνθεί ο συνδυασμό ε, οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Τι απαιτούμε λοιπόν. Πρέπει να υπάρχει πάντα μια επιλογή πολιτικής στα θέματα αυτά. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που ακολουθούμε τα τελευταία 20 χρόνια. Θα πρέπει να αλλάξουμε πολιτική και να έχουμε πιο συνεπή προσέγγιση, πιο συνεκτική προσέγγιση. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε το πρότυπο του εργαζομένου να είναι ένας εργαζομένος ο οποίος επίσης ε, να ε, φροντίζει την οικογένειά του. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι δυνατές ε, οι ευέλικτες ρυθμίσεις. Πρέπει να έχουμε ευέλικτες αδιαδρομίες, δηλαδή που να περιλαμβάνουν περιόδους ε, υψηλής ε, δραστηριότητας ε, και περιόδους πιο ήσυχες. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχα μια συζήτηση με γυναίκες που εργάζονται σε πανεπιστήμιο, που μπορεί να μην είναι η πρωταρχική ομάδα στόχος μας. Μας εξήγησαν όμως πόσο δύσκολο είναι να συνδυάσουν τις οικογενειακές υποχρεώσεις με την σταδιοδρομία σε πανεπιστημιακό επίπεδο, διότι δεν είναι τόσο απλή η εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους όσο είναι σε μια επιχείρηση. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε περισσότερο στις κοινωνικές υποδομές. Γι' αυτό επικρότησαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ε, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, νέα πρότυπα, διότι στις πολιτικές αυτές πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τα στερεότυπα που υπάρχουν. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τα οικογενειακά μοτίβα, να δούμε και να λάβουμε υπόψη μας τις διάφορες μορφές οικογένειας που υπάρχουν. Θα πρέπει να εξετάσουμε και το ρόλο των ανδρών και θα πρέπει να εργαστούμε παράλληλα πάνω στα πρότυπά μας. Μπορώ να σας παραπέμψω στη συζήτηση που είχαμε πάνω στο θέμα αυτό όταν διαπραγματευτήκαμε την αναθεώρηση της ρύθμισης για την γονεακή άδεια. Το θέμα δεν ήταν ότι οι, εργα... εργοδότες και οι εργαζόμενοι είχαν διαφορετικά πρότυπα ε, για την οικογένεια. Το θέμα είναι ότι υπήρχαν πολιτικές διαφορές ε, ε, σχετικά με το τι θεωρείται οικογένεια σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν βλέπετε τον οδηγό μας σχετικά με το πώς μπορεί να εφαρμοστεί η οδηγία, η αναθεωρημένη οδηγία για τις γωνιακές άδειες. Και στην ε, τελευταία μου διαφάνεια επανέρχομαι στα αιτήματά μας ε, που είναι αιτήματα άμεσα τα οποία σχετίζονται με την κρίση. Δεν ε, θα σας εκπλήξει ότι δεν στηρίζουμε τα μέτρα λιτότητας που έχουν επιβληθεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε επενδύσεις και υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες. Θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα θέματα που σχετίζονται με την οικονομική διακυβέρνηση. Στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ε, ε, αγνοείται σε μεγάλο βαθμό η ισότητα των φύλων και συνεργαζόμαστε με το Κοινοβούλιο για να αναθεωρήσουμε την οδηγία για την ψαλίδα στις αμοιβέ ανδρών και γυναικών. Υπάρχει μεγάλη επιφύλαξη από πλευρά των κρατών μελών να εξετάσουν το θέμα αυτό. Εμείς είμαστε υπέρ και μιας πατρικής άδεια. Πρέπει να ομολογήσω ότι όταν συζητήσαμε τότε το θέμα αυτό με το Κοινοβούλιο, συναντήσαμε κάποιες δυσκολίες ε, σχετικά με το αν θα πρέπει να συμπεριληφθεί η πατρική άδεια στην ε, οδηγία για την άδεια κοίησης και την μητρική άδεια. Ξέρουμε ότι η οδηγία αυτή έχει κολλήσει στα σιρτάρια της Κομισιόν. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις οι οποίες δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα επειδή υπάρχει ακόμα το θέμα πώς θα πρέπει να προωθηθεί η προστασία της μητρότητας. Τέλος, ε, ελπίζω οι άλλοι να μην έχουν τι ίδιες τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζω εγώ. Θέλουμε να φροντίσουμε να επιτευχθούν οι στόχοι τη Βαρκελόνη, ε, δηλαδή ε, δηλαδή να υπάρχουν διευκολύνσεις για τη φροντίδα των παιδιών σε όλη την Ευρώπη να μην περικοπούν λόγω τη λιτότητα. Νομίζω ότι περιορίστηκα στα 10 λεπτά. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Τώρα η Κωνσταντίνα Δαβάκη που είναι ερευνήτρια από το London School of Economics και θα είναι η δεύτερη μας ομιλήτρια που σε διάφορες ευκαιρίες είχε ξανά στην Επιτροπή μας και είχε μιλήσει για θέματα όπως γονική άδεια, Η κυρία Δαβάκη είναι Research Fellow στο LSE. Ετοίμασε μία θέση για το ρόλο των γυναικών στην αγορά εργασίας και την οικογένεια, συγκριτική προσέγγιση πολιτική στη Γερμανία και την Ελλάδα. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Okay. Well, Σας ευχαριστώ που με καλέσατε και μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για ένα τόσο συναρπαστικό θέμα που μας επηρεάζει όλες. Βεβαίως σε δέκα λεπτά μόνο κάποιες ιδέες μπορώ να δώσω γιατί νόμιζα ότι η συνεισφορά μου θα έπρεπε να ήταν να συνδέσω ιδέες, γιατί οι συνάδελφοι εδώ έκαναν πολύ καλή δουλειά παρουσιάζοντας μια στατιστικών στοιχείων. Και εσείς γνωρίζετε καλύτερη νομοθεσία από ότι εμείς. Ξεκινώ με το τι θεωρούμε κατά βάση ως ισορροπία εργασίας οικογένειας. Η ικανότητα να συνδυάσει κανείς τη δουλειά και την οικογένεια και επαγγελματικά και οικιακά. Ωστόσο πρέπει να διευρύνουμε το φάσμα αυτό συμπεριλαμβάνοντας όλες τις σύγχρονες ρυθμίσεις στην, στην οικογένεια ε, που είναι μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με παιδιά, οικογένειες ε, ζευγαριών του ιδίου φίλου κλπ. Και να έχουμε μία όσο πιο αντιπροσωπευτική κατάσταση μπορούμε θρησκευτικών ε, ομάδων, κοινωνικών ομάδων, κοινωνικών τάξεων και όχι την παραδοσιακή σχέση οικογένειας ενός λευκού ετεροφιλόφιλου ζευγαριού. Περιλαμβάνει λοιπόν το δικαίωμα μείωσης ε, των ορών εργασίας και την, το δικαίωμα στην γονική άδεια. Η συνάδελφος κυρία Μένεκ το κάλυψε αυτό, δεν θα μείνω στο θέμα αυτό. Αυτό που θα σας πω, που πιστεύω ότι είναι χρήσιμο, είναι πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ορισμούς των λειτουργημάτων που να επηρεάζουν το άτομο και την ευημερία μας. Θέλουμε τα άτομα να μπορούν να επιλέξουν τη μορφή ζωής που θεωρούν σημαντική, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο δουλειά και φροντίδα της οικογένειας, είναι μια πολυδιάστατη εμπειρία που περιλαμβάνει δουλειά, αναψυχή, εκπαίδευση, κοινωνική δέσμευση, διασκέδαση και οικογένεια. Ευτυχία, αυτοεκτίμηση, αυτοσεβασμό, ικανοποίηση από τη δουλειά. Αυτή η ευελιξία είναι κρίσιμη για να μπορέσουμε να κουμαντάρουμε αυτές τις δύο, αυτά τα δύο πλαίσια, τις δύο δομές ζωής, αλλά η πολλή ευελιξία μπορεί να μπλέξει τη δημόσια σφαίρα από την ιδιωτική σφαίρα. Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε μία σωστή κατανομή αμοιβόμενης και μη αμοιβόμενης δουλειά σαν δρόμο για τη μείωση των ενισοτήτων ε, μεταξύ φύλου στην επαγγελματική δραστηριότητα. Η ισορροπία λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβουμε πως ε, αυτό που και η κυρία Μένε ανέφερε, ότι δηλαδή είναι σημαντικό να αδράξουμε τις διάφορες φάσεις της ζωής του καθενός μας και ότι αυτό είναι μια διαδικασία δυναμική, όχι στατική ότι είναι μια κατάσταση ε, μεταβατική. Σήμερα μπορεί να είσαι ευχαριστημένη και παντρεμένη. Αύριο το πρωί θα χρησιμοποιήσω έναν όρο του Ζίκμουντ Μπάουμαντ. Μπορεί να είσαι σε άλλη κατάσταση. Άνεργος, διαζευμένος, μητέρα, μητέρα με παιδί χωρίς σύζυγο. Τα πάντα είναι σχετικά στη ζωή. Και πρέπει να αναφέρουμε ότι η μέρημνα σε έναν ε, γυράσκοντα πληθυσμό περιλαμβάνει και άλλες διαστάσεις πέραν της ε, ανατροφής των παιδιών. Και εκεί πρέπει να λάβουμε υπόψη την ευελιξία λοιπόν. Χρειαζόμαστε κοινωνιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να αντικατοπτρίζουμε την ε, διαφορετικότητα των κοινωνιών μας. Μια διατομεακή προσέγγιση είναι χρήσιμη γιατί επιτρέπει να καταλάβουμε πώς ε, συνδιαλέγουμε την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή αλλά και το πόσο διαφορετικές είναι οι καταστάσεις του καθενός μας. Αυτό που επίσης χρειάζεται είναι η αύξηση της επίγνωσης μεταξύ των γονέων σχετικά με το τι δικαιούνται και πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματα αυτά. Και σας λέω εδώ κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό το εισήγαγαν ο Χόψον και ο Τάκαρ σε μια ενδιαφέρουσα μελέτη όπου σύγκριναν τη χρήση των δικαιωμάτων των ε, επιδομάτων στην Ουγγαρία και την Σουηδία χρησιμοποίησαν τρεις ομάδες παραγόντων. Τον θεσμικό, επίπεδο πολιτικής, δικαιώματα, υπηρεσίες, επιδόματα, ποιότητα υπηρεσιών, συλλογική, συ, συ, διαπραγμάτευση και ατομικούς παράγοντες. Φύλλο, εθνική καταγωγή, πρόσβαση στους πόρους, ανθρώπινο κεφάλαιο, θέση στην κοινωνία και κοινωνιακούς παράγοντες. Κοινότητα, δημόσιου δημόσιος λόγος και κοινωνικά κινήματα. Μια χρήσιμη ένα χρήσιμο διάγραμμα που βλέπετε εδώ έχει στόχο να σας πει πως όλοι αυτοί οι παράγοντες συνδέονται μεταξύ τους και οδηγούν από την ύπαρξη των δικαιωμάτων στην υλοποίηση των δικαιωμάτων από τον ε, δρόντα το άτομο στη συγκεκριμένη περίπτωση μέχρι την έννοια του δικαιώματος που διεκδίκησε. Αυτό δείχνει ότι στους άξονες που συνδέονται μεταξύ τους εδώ λείπει κάτι. Μπλοκάρεται η υλοποίηση των δικαιωμάτων. Δηλαδή, αν η κουλτούρα του χώρου εργασίας δεν παρέχει πολλές ε, μεγάλο βαθμό ανεκτικότητας τα δικαιώματα χρησιμοποιούνται πολύ λιγότερο. Επίσης, ζούμε μεσούσεις οικονομικής κρίσεως. Θα αναφέρω λοιπόν εντάχει ορισμένες επιπτώσεις στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Πρώτον, ε, η διάσταση φύλου στην καταγραφή της ανεργίας και της φτώχειας. Ε, στα... Υπάρχει πόλωση και στα δύο άκρα της κλίμακας. Διευρύνονται οι ανισότητες εισοδήματο. Το γεγονός ότι επιδεινώθηκε η κατάσταση των ανδρών δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρόοδος στην ισότητα των φύλων. Δεύτερον, οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο, ξέρουμε γιατί ήδη αναφέρθηκε, κυρίως διότι υπερεκπροσωπούνται στο δημόσιο σε πολλές χώρες, χώρες που έχουν υποστεί τις επιπτώσεις της κρίσης και που μείωσαν σημαντικά τον αριθμό των υπαλλήλων του δημοσίου και άρα και των ε, γυναικών εργαζομένων εκεί. Επίσης, υπερεκπροσωπούνται σε όλες ε, τις δραστηριότητες ε, οικογενεια... μέρημνας οικογένειας. Αυτό το θέμα το έχετε συζητήσει σε τρεις ακροάσεις ήδη και σε όλες τις χώρες που αντιμετωπίζουν κρίση οι πρόνοια, οι προνοιακές πολιτικές έχουν πληγεί περισσότερο. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι η πρόνοια έχει μεγάλη κοινωνική αξία αλλά μικρή αγοραστική αξία. Κάτι επίσης ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με τις πρόσφατες μελέτες η συμπεριφορά των γεγών στην αγορά εργασίας ε, μέσα στην κρίση άλλαξε. Βλέπουμε λιγότερες γυναίκες να είναι έτοιμες να βρουν μερικής απασχόλησης δουλειές. Κάτι που είναι παρηγορητικό. Ωστόσο, και πάλι, αυτό δεν υπάρχει γιατί υπάρχουν άλλες θέσεις, μαξιλα, άλλες θέσεις εργασίας μαξιλαράκια που καλύπτονται τώρα από νεότερους ή μετανάστες. Αυξήθηκε ταυτόχρονα η φροντίδα της οικογένειας με επίπτωση, αρνητική επίπτωση στη γυναίκα. Όλα αυτά οδηγούν στη δυνατότητα ωστόσο να ελπίσουμε για ριζικέ αλλαγέ. Και αυτό γιατί είμαι αισιόδοξη. Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν τώρα για την ισότητα των φύλων. Ε, η μείωση του αριθμού των εργαζομένων στο δημόσιο και η μείωση των μισθών είναι ο κύριος κίνδυνος. Άρα πρέπει να υπάρξουν ε, γρήγορα ρυθμιστικά μέτρα που θα εξασφαλίσουν ότι η, το κέρδος της παραγωγικότητας θα διανεμηθεί το συντομότερο δυνατό. Όρια κριτηρίων επιλεξιμότητας προφανώς δεν επηρεάζονται όλα τα κράτη-μέλη, ε, δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη την ίδια εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Ένα άλλο θέμα είναι ότι το mainstreaming φύλου δεν εφαρμόζεται ως απάντηση στην κρίση. Η οικονομική, η δημοσιονομική εξυγίνηση, οι προσπάθειες ανάκαμψης δεν εξετάζονται από την οπτική της επίπτωσης στην ισότητα φύλου. Και εδώ τίθεται το ζήτημα του πώς αντιμετωπίζουμε τα κοινωνικά προβλήματα γενικότερα. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε απομονώνοντας στους τέσσερις αυτούς παράγοντες. οικονομία και τον ε, κοινωνικό τομέα και τον πολιτικό τομέα. Και γιατί σας τα δείχνω όλα αυτά. Γιατί έχω την άποψη ότι αν δεν δούμε τις προνοιακές πολιτικές με έναν ολιστικό τρόπο, θα καταλήξουμε σε λάθος συμπεράσματα. Διότι οι περικοπές στην μία πλευρά οδηγούν σε αύξηση δαπανών σε άλλο τομέα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ανεργία. Η αύξηση στην ανεργία επηρεάζει διάφορες κατηγορίες επαγγελμάτων και κοινωνικές τάξεις. Μετά υπάρχει το θέμα της στέγασης. Και πώς επηρεάζονται η στέγαση και η υγεία. Έχουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι η υγεία, ιδίως η ψυχική υγεία, υγεία μειώνεται, επιδεινώνεται στην Ευρώπη. 30 εκατομμύρια άτομα έχουν κατάθλιψη στην Ευρώπη τώρα. Δεν θα πω περισσότερο σε λεπτομέρειες, αλλά να τονίσω την σχέση μεταξύ πολιτικών και συμπεριφορών, διότι οι συμπεριφορές επηρεάζονται αλλά και διαμορφώνονται από τις πολιτικές. Τώρα θα τελειώσω με τις νέες τάσεις και ανησυχίες πολιτικής. Πρώτον, αύξηση δυσαρέσκειας των πολιτών της Ένωσης έναντι των κυβερνώντων εν γέννη. Ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, επιστροφή σε ένα στυλ ζωής λιγότερο καταναλωτικό, μιλώ για τις ε, χώρες που επλήγησαν από την κρίση, αύξηση της κατάθλιψης και αύξηση της βίας κατά των γυναικών και των μεταναστών. Και ρατσισμό. Υπό το φως της Ευρώπης 2020, ε, η ύφεση υπονομή μεύει τις, τα επιτεύγματα για την ισότητα των γυναικών και τα μέτρα για την ισότητα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται και πριν και κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους. Ο μόνος δρόμος μπροστά είναι η γονική άδεια. Δεν πρέπει να υπάρχουν περικοπές στις ρυθμίσεις μητρικής άδεια για να ξεκινήσουν καλά τη ζωή τους τα παιδιά μας. Καλύτερα οδηγίες, όχι συστάσεις. Και επαναφορά θεσμών ισότητας ε, σε διάφορες χώρες που υπήρχαν αλλά οι αρμοδιότητές τους περιορίστηκαν ή ε, εξαφανίστηκαν. Και να σας δώσω και κάποιες παραθέσεις που βρήκα ενδιαφέρουσες. Είμαστε ευτυχείς να ζούμε στην Ευρώπη που γέννησε τη δημοκρατία και το κράτος ε, πρόνοιας. Αυτό είναι αξία που πρέπει να διαφυλάξουμε. Ας ακούσουμε τη φωνή του λαού μας. Ας καταλάβουμε την ματέωσή τους. Ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος. Στη ζωή υπάρχουν ατυχήματα και ανθρωπογενείς καταστροφές. Εάν μπορέσουμε να περιορίσουμε ή να αποφύγουμε το τελευταίο, είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Η ανάπτυξη είναι σημαντική, αλλά με τι κόστος. Τελειώνω λέγοντας ότι οι ανθρωπογενείς καταστροφές αποδείχθηκε ότι μπορούν να σωθούν. Οι, τράπεζες, οι κυβερνήσεις έδειξαν ότι μπορούν να σώσουν τις τράπεζες, μπορεί να σώσουν και γενιές ανθρώπων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καδαβάκη. Τελευταίος ομιλήτρια σε αυτό το γύρο, Άνια Σπανεφάριαν, που την καλώ τώρα να έρθει στο βήμα. Έχει 15 ετή εμπειρία σε θέμα κοινωνικών ερευνών στην Ευρώπη. Δουλεύει στο Eurofound και είναι υπεύθυνη για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τις συνθήκες εργασίας. Αρμόδια δε για θέματα φύλου. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Δέκα λεπτά κι εσείς. Έχουμε ήδη δεκα, δεκάλεπτη καθυστέρηση. Περιμένουμε να δουλέψει το μηχάνημα λίγο. Θα μιλήσω στα γαλλικά, γι' αυτό αν θέλετε βάλτε ακουστικά. a little problem with the computer. Yes. Voilà, excusez-moi pour... Με συγχωρείτε για αυτή τη μικρή καθυστέρηση, τέλο πάντων. Λέγομαι Ανιές Παραντεριού και είμαι Senior Program Manager στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα. Εκεί σε συνεργασία με κυβερνήσεις και κοινωνικούς εταίρους προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής και εργασίας. Αυτό. Λοιπόν, θα θέσω τα ίδια ερωτήματα με τις προηγούμενες, αλλά θα δώσω και αριθμούς και ελπίζω να μπορέσετε να τους δείτε στην οθόνη. Αλλιώς Έχουμε την έκθεση εδώ και τυπωμένη και μπορείτε να τη διαβάσετε. Εξηγεί ακόμη καλύτερα αυτά που θα έλεγα. Καταρχήν, θέλουμε να εξετάσουμε το θέμα της εξορρόπησης δουλειάς και οικογενειακής ζωής. Όλοι συμφωνούμε στο στόχο, αλλά δεν είμαστε όλοι σίγουροι αν καταλαβαίνουμε τα ίδια πράγματα. Η εξισορρόπηση λοιπόν αυτή μπορεί να εξεταστεί με βάση τον τρόπο που οργανώνει ο καθένας τη δουλειά και την εργασία του κάθε μέρα. Εδώ η γραφική παράσταση είναι η απάντηση στο ερώτημα έχετε καταφέρει την εξισορρόπηση. Συνολικά 80% λένε ότι την έχουν πετύχει. Στις λεπτομέρειες όμως βλέπουμε ότι οι άντρες κυρίως και μάλιστα οι νέοι πατέρες είναι οι πιο δυσαρεστημένοι για αυτό το θέμα της εξισορρόπησης εργασίας και οικογενειακής ζωής. Θα μπορούσε κανείς να το δει με βάση όλη την καριέρα κάποιου ανθρώπου και εδώ βλέπουμε ότι ο χρόνος εργασίας ανά άνθρωπο Για τους άντρες είναι 37 περίπου χρόνια κατά μέσο όρο και κατά 8 χρόνια μεγαλύτερη από ότι ο χρόνος εργασίας των γυναικών. Για να καταλάβει κανείς καλύτερα πώς εξισορροπείται η οικογενειακή, η ιδιωτική με τη ζωή με την εργασία. Χρησιμοποίησα και εγώ τρεις κύκλους, όχι ακριβώς τους ίδιους με εσάς, αλλά πρέπει να δούμε και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, όπως τους παιδικούς σταθμούς, τα σχολεία κλπ. Γιατί αυτά είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί κανείς να εγγράψει την επαγγελματική του δραστηριότητα, επίσης την αγορά εργασίας που είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας και η άνηση μεταχείριση των φύλων στην αγορά εργασίας. Γιατί διαπιστώνουμε ότι μπορούμε και αυτό να το δούμε με διαφορετικούς τρόπους, οι δυνατότητες δηλαδή που έχουμε να κάνουμε επιλογές για την εξισορρόπηση οικογενειακής ζωής και εργασίας. Εξαρτάται από το αν κανείς έχει σύντροφο, αν έχει και πόσα παιδιά κτλ. Βέβαια είναι διαφορετικά και τα καθήκοντα ανδρών και γυναικών. Αν θέλουμε λοιπόν να βελτιωθεί η εξισορρόπηση, δεν υπάρχει μία και μόνη πολιτική που πρέπει να εφαρμόσουμε, αλλά πολλές. Και μετά βέβαια τίθεται το ερώτημα εάν η πολιτική που εφαρμόζουμε είναι ολιστική ή συνεπής. Σημαντικό και αυτό το ερώτημα. Έχουμε ιδέες αλλά δεν έχουμε πραγματικά παραδείγματα. Θα σας δείξω τώρα τι γίνεται με τον κύκλο ζωής. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δει κανείς την άνηση μεταχείριση. Δεν έχουν κάνει όλοι τις ίδιες σπουδέ και γι' αυτό δεν κάνουν και την ίδια δουλειά. Υπάρχουν τα πιο συνήθιοι επαγγέλματα, 76% δηλαδή των επαγγελμάτων δείχνουν ότι οι 20 ομάδες που τα αποτελούν από τις 20 ομάδες που τα αποτελούν μόνο 5 είναι μικτές. Είναι εξαίρεση να δουλεύει κανείς σε ένα μεικτό περιβάλλον. Συνήθως οι άντρες δουλεύουν με άντρες και οι γυναίκες με γυναίκες και πολύ λιγότερο συχνά σε μεικτό περιβάλλον. Άλλο παράδειγμα της άνησης μεταχείρισης είναι πρώτον ότι υπάρχουν πολύ λιγότερες γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις. Δεύτερον, ακόμη και όταν είναι διευθύντριες, ε, διοικούν συνήθως μικρότερες ομάδες, περισσότερο με μερική εργασία και σε τομείς με χαμηλότερους μισθούς. Ακόμα και όταν οι γυναίκες λοιπόν φτάνουν σε διοικητικές θέσεις, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από των ανδρών. Άλλο παράδειγμα, έχει διαλέξει κανείς ένα επάγγελμα, ας πούμε όπου υπάρχουν περισσότερες γυναίκες, είναι ή δεν είναι σε διοικητική θέση και προστίθεται εδώ ένα επίπεδο. Σε 20% των περιπτώσεων σε μια επιχείρηση μεικτή, μεικτής απασχόλησης, μόνο υπάρχει αυτός ο μικτός χαρακτήρας. Αυτά όλα τα επίπεδα διαφορετικής μεταχείρισης μπορούν και να συνδυαστούν. Πάντως ο μικτός χαρακτήρας είναι εξαίρεση ακόμα. Όταν είναι μεικτή εργασία και άντρες και γυναίκες μαζί, τα αποτελέσματα είναι θετικότερα. Τώρα περνάω στο ότι έχει κανείς το επάγγελμά του στην επιχείρησή του, τι τύπο εργασίας κάνει και ποια είναι η ποιότητα της εργασίας του. Αυτό μας απασχολεί πολύ στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα. Δημιουργήσαμε πολλούς δείκτες για την ποιότητα εργασίας και θα σας παρουσιάσω τώρα τέσσερις από τους κύριους δείκτες ανάλογα με το... τη φάση της εργασιακής ζωής. Η μία είναι στην αρχή της απασχόλησης, η δεύτερη ε, μέχρι 45 ετών, μετά παντρεμένη με ή χωρίς παιδιά και μετά η τελευταία φάση όπου έχουν φύγει τα παιδιά. Τι βλέπουμε λοιπόν ότι διαφέρουν τα πράγματα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ίσως είναι κοινοτόπο κοινότοπο αλλά το ροζ αντιπροσωπεύει τις γυναίκες εδώ και το μπλε τους άντρες. Και βλέπουμε ως προς την ποιότητα της εργασίας ότι οι γυναίκες γενικά έχουν μεγαλύτερη ποιότητα εργασίας από τους άντρες αλλά οι συνδυασμοί είναι ενδιαφέροντες. Οι γυναίκες ε, δουλεύουν πολύ λιγότερο συχνά τη νύχτα και λιγότερες ώρες. Πολύ περισσότερο όμως σε μερική εργασία και αυτό θέτει πρόβλημα εισοδημάτων και έχουν πολύ λιγότερες δυνατότητες επιλογής και προσαρμογής των ωραρίων τους. Ένας νέος δείκτης είναι αν μπορώ να ζητήσω από τον εργοδότη μου μια-δυο ώρες να φύγω για το γιατρό ή για άλλες δουλειές και πολύ περισσότεροι άντρες έχουν αυτή τη δυνατότητα από ότι γυναίκες. Καλύτερη ποιότητα λοιπόν του χρόνου εργασίας των ανδρών από τη μία, ναι, ως προς την υγεία, αλλά δεν υπάρχουν οι ίδιες δυνατότητες και ευκολίες. Άλλο θέμα, οι προοπτικές για το μέλλον σε ποιο βαθμό μπορεί κανείς να αναμένει ότι θα εξελιχθεί η καριέρα του ή απλώς και ότι θα διατηρήσει την εργασία του. Εδώ βλέπουμε ότι από τη στιγμή που υπάρχουν παιδιά οι προοπτικές μειώνονται. Δεν τα θεωρώ σε αιτία και, αιτία και αποτέλεσμα, αλλά είναι δύσκολο να συνδυάσει κανείς εδώ την οικογένεια με την εργασία εάν δεν υπάρχει ασφάλεια, κοινωνική ασφάλεια. Τρίτος παράγοντας η ίδια η ποιότητα εργασίας. Εκτίθεται κανείς σε φυσικούς κινδύνους ή σε κοινωνικό περιβάλλον που δεν το ανέχεται ή σε πράξεις βίας κλπ και σε ποιο βαθμό μπορούμε εμείς να είμαστε χρήσιμοι. Εδώ βλέπουμε ότι οι γυναίκες έχουν πιο υψηλή ποιότητα εργασίας με αυτά τα κριτήρια γιατί εκτίθενται λιγότερο σε φυσικούς κινδύνους. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές διαφορές και υπάρχει και το θέμα των μισθών βέβαια δεν μιλάω πολύ γι' αυτό αλλά η μερική εργασία, τα ανισότητες ε, στη μισθοδότηση μεταξύ ανδρών και γυναικών, όλα αυτά αφορούν επίσης το, την ποιότητα ζωής και τελικά οι συντάξει ας πούμε είναι πάρα πολύ διαφορετικές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αν τα εξετάσουμε με το εύρος ολόκληρου κύκλου ζωής είναι τεράστια η διαφορά και η ισότητα των φύλων και ως προς αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Το μεγάλο θέμα, η μεγάλη διαφορά είναι το θέμα του χρόνου. Πόσο χρόνο δαπανά κανείς κάθε μέρα στην εργασία του και στις μεταφορές καθώς και για την ανατροφή των παιδιών. Οι γυναίκες συνεχίζουν να φέρουν το μεγαλύτερο βάρος για τα οικιακά και τα παιδιά. Προσπαθήσαμε να υπολογίσουμε τις 68 ώρες που αντιπροσωπεύουν μία εβδομάδα και είδαμε ότι οι άντρες εργάζονται περισσότερο από τις γυναίκες αλλά αν συνδυάσουμε τη μισθωτή εργασία με την αμίσθωτη οι γυναίκες εργάζονται περισσότερο. Οι γυναίκες πρέπει να αντιμετωπίσουν και άλλα καθήκοντα από ότι οι άντρες που ασχολούνται απλώς με την μισθωτή τους εργασία, αμοιβόμενη εργασία. Αν κοιτάξει κανείς όμως το θέμα της ευημερία, βλέπει ότι οι άντρες θεωρούν ότι έχουν μεγαλύτερη ευημερία και ότι δεν μειώνεται πουθενά το χάσμα. Συμπαρασματικά λοιπόν, αν θέλουμε να βελτιωθεί, όχι μάλλον όχι, αν θέλουμε να βγει η Ευρώπη από την κρίση πρέπει να δούμε το θέμα της εξισορρόπησης εργασίας με οικογενειακή ζωή. Βεβαίω είναι πολύπλοκο το πρόβλημα γιατί όπως είδατε υπάρχουν πολλά επίπεδα που πρέπει να συνδυαστούν. Γι' αυτό χρειάζεται ολόκληρη σειρά προγραμμάτων και πολιτικών. Πρέπει να καταπολεμηθούν οι ανισότητες και πρέπει και να μειωθεί ο μικρός και ο μεγάλος χρόνος μερικής απασχόλησης. Οι άντρες και οι γυναίκες θέλουν να εργάζονται τον ίδιο χρόνο. Ως προς την ποιότητα της εργασίας και της απασχόλησης πρέπει αυτοί που μπαίνουν στην αγορά εργασίας να έχουν ήδη από την αρχή εισοδήματα επαρκή για να επιβιώσουν και καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής να μπορούν να αντιμετωπίσουν διάφορα απρόβλεπτα ατυχήματα κλπ. Και να έχουν πόρους όχι μόνο οικονομικούς αλλά και το πώς θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τις δεξιότητές τους. Πρέπει λοιπόν η προσέγγιση να είναι ευρεία και σταματώ εδώ. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, agnes Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα φτάσαμε στο τέλος του πρώτου γύρου και αρχίζουν οι ερωταπαντήσεις των συναδέλφων. Έχω ήδη κάποιον που έχει ζητήσει το λόγο. Η κυρία Μόρβάη έχει το λόγο. Θα μιλήσω ουγγαρέζικα. Παροδία είναι αυτό μια κοινή σύνοδος δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών και μια ακρόαση στην οποία μετέχουν μη κυβερνικές οργανώσεις. Κανονικά θα έπρεπε να έχουμε δηλαδή εδώ 80 βουλευτές παρόντες. 8 είναι παρόντες. Κοινή συνεδρίαση δύο επιτροπών που ενδιαφέρει 8 ευρωβουλευτές. ένα θέμα που είναι σημαντικό. Την ε, ισορροπία οικογενειακή και ζωή ζωής ένα κρίσιμο θέμα για το μέλλον της Ευρώπης. Επίσης, είναι μια παροδία του ότι ε, πράγματα σημαντικά σε μια μικρή πόλη δεν μπορούν να ενδιαφέρουν το κοινοβούλιο. Μιλάμε για ισότητα ανδρών γυναικών γενικά χωρίς να καταλαβαίνουμε τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις γυναίκες στις περιοχές της περιφέρειας και τις γυναίκες στις κεντρικές χώρες της Ευρώπης. Το ίδιο πρόβλημα εμφανίζουν πάρα πολλοί πολιτικοί και ειδικοί. Μιλούν για ένα ζήτημα χωρίς να διακρίνουν ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Υπάρχουν βασικές διαφορές ανάμεσα στο πώς ένας άντρας και μια γυναίκα καταλαβαίνει το να συντεριάξει οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Αλλά και εδώ το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε γενικεύουμε. Γιατί γενικεύουμε, γιατί το κοινοβούλιο λειτουργεί με τον τρόπο αυτό στην Ουγγαρία, νέο κράτος μέλος, σε μετακομμουνιστική περίοδο, οι γυναίκες υφίστανται μία σύγχρονη δουλεία. Έχουν μικρή συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Και ρωτώ την εκπρόσωπο των συνδικάτων, τι ξέρετε για την κατάσταση των γυναικών στην Ανατολική Ευρώπη. Ξέρετε ότι είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης από δυτικές πολυεθνικές εταιρείες που τιμωρούν τη συμμετοχή τους σε εργατικά συνδικάτα. Αυτό έχει επιπτώσεις σε γυναίκες ε, που είναι πιο ευάλωτες από ό,τι άνδρες συχνά είναι χρεωμένες, πρέπει να πληρώσουν δάνεια. Δεν θα μιλήσω περισσότερο για το θέμα αυτό, αλλά οι γυναίκες σε κάποιες καταστάσεις βρίσκονται σε πολύ ευάλωτη θέση γιατί και επιπλέον δεν μπορούν να μπουν και σε συνδικάτο γιατί δεν τις απέλυαν. Η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Ρωτώ λοιπόν, τι ξέρετε για την κατάσταση των γυναικών στην Ανατολική Ευρώπη στον τομέα της συνδικαλιστικής, ε, του δικαιώματος του συνεταιρίζεστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ οι ερωτήσεις σας να είναι σύντομες, δεν θέλουμε μακροσκελείς παρεμβάσεις. Η συνάδελφος Κορνέλης έχει το λόγο. ευχαριστώ. πολύ κυρία Πρόεδρε. Η παρουσία 8 βουλευτών είναι πολύ χαμηλή βέβαια, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι για τις ακροάσεις μας είναι συνήθως ακόμα λιγότεροι. Εδώ φαίνεται υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι συνήθως. Λοιπόν, θυμάμαι πολύ καλά μια κρόαση πριν από 1,5 χρόνο όπου υπήρχε ένας Νορβηγός ομιλητής και είπε στην Νορβηγία η εξισορρόπηση ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής θεωρείται σαν επένδυση στην οικονομία μας και θυμάμαι ότι ζήλεψα πάρα πολύ διότι εγώ ζω στην Ολλανδία και εκεί σίγουρα δεν το βλέπουν έτσι. Δύο μέρες ας πούμε γονικής αδείας τη μία για να γιορτάσουν και τη δεύτερη για να εγγράψουν το παιδί τους στα Μητρώα. Δύο μόνο μέρες και δεν άλλαξε από τότε. Γενικά οι υπηρεσίες για τα παιδιά είναι πολύ χαμηλής ποιότητας. Δεν υπάρχει δηλαδή στην Ολλανδία η αντίληψη ότι είναι όλα αυτά επένδυση και στην οικονομία. Αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους του 2020, να μειώσουμε την ανέχεια, που πλήττει περισσότερο τις γυναίκες από τους άντρες, να αυξήσουμε την απασχόληση, γιατί οι γυναίκες είναι ο μεγαλύτερος ανεκμετάλλευτος πόρος για την απασχόληση. Θα, αν θέλουμε λοιπόν να τα πετύχουμε όλα αυτά, μας έχετε δώσει πολύ σημαντικές πληροφορίες και εργαλεία για να ζητήσουμε από την Κομισιόν μια συνολική πολιτική, όχι κατακαιρματισμένα τα θέματα, τη γονική άδεια, τους στόχους της Βαρκελόνης κλπ. Όλα τα βλέπουμε κατακαιρματισμένα και σαν θέματα που αφορούν μόνο τις γυναίκες ενώ πρέπει να υπάρξει μια συνολική πολιτική ζωτική για το μέλλον ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικονομίας σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτά τα εργαλεία που μας διαθέσατε, γιατί είναι σημαντικά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος, κυρία Μπαλτατσίνο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι συντομότατη. Θέλω να ρωτήσω αν η εξισορρόπηση ιδιωτικής και επαγγελματική ζωής γιατί μάλλον περιορίζεται μόνο στην τεκνογονία. Εδώ υπάρχουν δημογραφικές αλλαγές. Υπάρχουν μητέρες που είναι και επαγγελματίες αλλά και γυναίκες που πρέπει να απασχοληθούν όχι μόνο με τα παιδιά τους αλλά και με τους γονείς τους. Τι θα κάνουν. Μιλάμε βέβαια για τα παιδιά, αλλά δεν μιλάμε ποτέ για τους γονείς που είναι ηλικιωμένοι και τα, και τα παιδιά τους δεν θέλουν να τα βάλουν σε γυροκομεία, θέλουν να τους φροντίσουν, αλλά αν έχουν κάποια δουλειά, αν είναι καθηγητές ας πούμε, τι θα κάνουν. Θα αφήσουν τους φοιτητάς των για να πάνε να ασχοληθούν με τους γονείς τους ή θα αφήσουν στο νοσοκομείο τη μητέρα τους διότι είναι, έχουν τη δουλειά τους, είναι ας πούμε μηχανικοί. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Γιατί υπάρχουν γυναίκες που δεν έχουν παιδιά, έχουν όμως γονείς. Δεν κάνουν όλες οι γυναίκες παιδιά. Καλό είναι που το λέμε και αυτό αλλά θα ήθελα το Κοινοβούλιο να μιλήσει και για τις γυναίκες που έχουν μια δουλειά και πρέπει να ασχοληθούν γενικότερα με την οικογένειά τους. Το σκεφτήκατε λοιπόν ποτέ, αυτό ερωτώ. Ευχαριστούμε πολύ. Απαντήσεις. Πρώτα, η κυρία Κλάουδια Μένε. Μετά για τη δεύτερη ερώτηση την κυρία Κορνέλ. Α, όχι, υπάρχει και άλλη ερώτηση Τη της κυρίας Λούλινγκ. Ευχαριστώ. Όχι ερώτηση. Απλά να σας πω ότι αυτό που άκουσα για τις εκδικήσεις με οδηγούν στο να Σκεφτώ, ξέρετε, τις ε, πάμπολες οδηγίες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ευτυχώς για την ισότητα ευκαιριών ανδρών και γυναικών. Από το 1975 έχουμε οδηγίες, 11 νομίζω τώρα, που ασχολούνται με το θέμα. Στην ουσία παραβιάζεται ανοιχτά σφύρας Προφανώς κάποιες μπορούν να βελτιωθούν. Αυτή για την άδεια μητρότητας, για παράδειγμα. ...άρα το Κοινοβούλιο έκανε εκεί το τεράστιο λάθος να περιλάβει ένα κείμενο που είχε τα πάντα μέσα. Με, απί, με απίθανες απαιτήσει με την οποία δεν ασχολήθηκε καμία προεδρία. Αν κάναμε μία λογική πρόταση, θα είχαμε άδεια μητρότητας, ελάχιστη άδεια μητρότητας σε όλη την Ένωση εδώ και δύο χρόνια. Μεγαλύτερη από ό,τι τώρα. Τώρα υπάρχουν 14 εβδομάδες. Η Επιτροπή είχε προτείνει 18. Τι κάναμε εμείς, προτείναμε 20 άδεια πατρότητας, όλα τα βάλαμε μέσα. Οι νόμοι πρέπει να μπορούν να εφαρμόζονται. Δεν βάζουμε λοιπόν τα πάντα. Έχουμε μια οδηγία για την ισότητα μισθών. Α την χρησιμοποιήσουμε. Αν την κάναμε τώρα, το 75 έγινε. Αν την κάναμε τώρα που είμαστε 28, δεν θα ήταν τόσο καλή όσο τώρα. Γιατί δεν εκμεταλλεύεστε αυτή την οδηγία. Εγώ στη χώρα μου το κάνω. Καταβλήθηκαν αναδρομικά εκατομμύρια σε γυναίκες, αλλά πρέπει να υπάρχει θάρρος. Και άλλωστε λέμε μη, υψηλότερη μισθή, η οδηγία μιλά το, για το άτομο, όχι το μέσο. Η οδηγία είναι για να ξέρεις ότι αν κάνεις ίδια δουλειά με αυτή που κάνει ένας άντρας και αντιμετωπίζεις διάκριση στην επιχείρησή σου ή στον τομέα σου ότι υπάρχει συλλογική σύμβαση πρέπει να διεκδικήσεις το δικαίωμά σου. Γιατί όχι. Δεν μπορώ να ακούω όλα αυτά, όλους αυτούς τους θρήνους. Ζητάμε πράγματα που υπάρχουν και δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει το θάρρος να το διεκδικήσουν. Για την γονική άδεια υπάρχει οδηγία. Τα κράτη-μέλη μπορούν να την ερμηνεύσουν όπως θέλουν, αλλά κάτι πρέπει να κάνουν. Στη χώρα μου ήταν ένας χρόνος και με πολύ καλή αμοιβή. Σε άλλες χώρες είναι κάτι άλλο. Αλλά αυτή είναι η επιλογή των χωρών. Το κοινοτικό κείμενο υπάρχει. Ναι, ναι, να σταματήσω. Με συγχωρείτε κιόλα. Ξέρετε, πιέζει ο χρόνος, γι' αυτό. Λυπάμαι. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για αυτό τα σημαντικά θέματα. Έχουμε πέντε λεπτά μόνο. Για τις απαντήσεις. Απαντήστε. Ξέρω ότι μπορείτε να απαντήσετε καλά σε λίγα λεπτά. Πέντε λεπτά και οι τρεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ένα λεπτό. Όσον αφορά τα συνδικαλιστικά δικαιώματα στην Ουγγαρία και τις πολυεθνικές, ε, θα πρέπει να επανέλθω. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση στην Ουγγαρία. Ε, έχετε και το σύστημα που γνωρίζουμε από την ε, Γερμανία. Ε, έχετε τα Συμβούλια της Επιχείρησης ε, και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσω τι γίνεται στον τομέα της λιανικής. Πάντως <coughs> γνωρίζουμε ότι οι πολυεθνικές συχνά παρενοχλούν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Δεν είναι όμως αποκλειστικά ουγγρικό φαινόμενο αυτό. Αν μπορούμε να ανταλλάξουμε email θα προσπαθήσω να επανέλθω. Οι ουγγρικές συνδικαλιστικές οργανώσεις προσπαθούν τώρα πια να εργάζονται πιο αποτελεσματικά και χρησιμοποιώντα και τι αρνητικέ εμπειρίε που έχουν τα τελευταία χρόνια. Ολοκληρωμένε στρατηγικέ. Ε, ναι, και εγώ ήθελα να σα μεταφέρω αυτό το μήνυμα. Είχαμε το παράδειγμα της ε, ε, γονεϊκής άδεια. Θα πρέπει να τα επαναξετάσουμε όλα αυτά και να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Πρόκειται για μια προσφορά από την ε, πλευρά μου, από την πλευρά των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Υπήρξαν κάποιε τριβέ ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και τι ε, οργανώσει γυναικών στο θέμα αυτό. Ίσως μπορούμε να αφήσουμε πίσω μα αυτέ τι αρνητικέ εμπειρίε. Ε, όσον αφορά το τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια εταιριών είχαμε καλύτερα εμπειρίες. Ίσως είναι χρήσιμο να επαναξετάσουμε τις εμπειρίες αυτές όταν θα εξετάσουμε τα νέα προγράμματα. Θα κλείσω εδώ. Ελπίζω να μην ξεπέρασα το ένα λεπτό. Ωραία. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι καλός κακό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να απαντήσει σε, όλες, σε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η εφαρμογή της όμως ε, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το κάθε κράτος μέλος. Πιθανότατα να πρέπει να εκλέξουμε τους ε, κατάλληλους πολιτικούς αν θέλουμε να προχωρήσουν κάποια ζητήματα. Ανέφερα την Ουγγαρία, όπως τη γνωρίζω εγώ. Και στην ε, Ουγγαρία ο κόσμος ένιωσε ότι οι άντρες δεν μπορούν καθόλου να ζητήσουν γονεακή ε, άδεια λόγω της κατάστασης στον εργασιακό χώρο. Υπάρχουν ε, όμως κάποια ελπιδοφόρα σήματα. Να επανέλθω στην κυρία που ρώτησε που έθεσε την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση σχετικά με τη φροντίδα των παιδιών. Ε, νομίζω ότι ανέφερα στην εισαγωγική μου παρέμβαση ότι θα πρέπει στο θέμα αυτό να συμπεριλάβουμε και τη φροντίδα των ηλικιωμένων, ε, οποιοδήποτε μορφής φροντίδα, όχι μόνο τη φροντίδα των παιδιών. Είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε αυτήν την οδό. Και όσον αφορά την κυρία που αποχώρησε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο για να πούμε γιατί κάποιοι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν το θάρρος να απαιτήσουν την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Πιθανότατα επειδή είναι φτωχοί, πιθανότατα επειδή είναι μετανάστες. Μερικές φορές μάλιστα είναι ε, παράνομα διαμένοντες. Νομίζω ότι κάλυψα τις ερωτήσεις που μου τέθηκαν. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, ναι, δεν είμαστε όλοι ίσοι. Υπάρχουν διάφορες ομάδες ανδρών και γυναικών που εκτίθενται σε διάφορες καταστάσεις ε, που ε, επηρεάζουν ε, την ισορροπία ανάμεσα στον οικογενειακό και επαγγελματικό βίο. Είναι λοιπόν θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης να αποφασίσουμε αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα γενικά ή αν θέλουμε να επικεντρωθούμε σε κάποιες ομάδες και το πώς θα ορίσουμε αυτές τις ομάδες. Είναι δύσκολο να βρούμε μια προσέγγιση που να ταιριάζει σε όλους λόγω αυτής της ποικιλομορφίας όσον αφορά το θέμα της φροντίδας των ηλικιωμένων. Όλοι ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, δεν το αναφέραμε. Υπάρχει και η λεγόμενη γενιά σάντουιτς ε, που ε, πρέπει να φροντίσει και την γενιά πριν και την επόμενη. Είναι λοιπόν ε, δύσκολο το θέμα αυτό και αφορά όχι μόνο τις γυναίκες. Αφορά και τους άντρες. Και γιατί οι άνθρωποι δεν ασκούν τα δικαιώματά τους. Έχουμε κάποια δικαιώματα, εξετάζοντα όμω τα δεδομένα, βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζονται τα δικαιώματα αυτά. Ίσως ε, να μπορέσουν να βοηθήσουν κάποια ε, συγκεκριμένα παραδείγματα. Αλλά υπάρχουν πολλοί παράγοντε ε, στην άσκηση δικαιωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο που διαδραματίζουν οι συνδικαλιστικέ οργανώσει. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα. Και ναι, όσον αφορά την ολοκληρωμένη στρατηγική, <laughs> ναι, θα το θέλαμε πάρα πολύ, θα σας ψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. E Ευχαριστώ. Κλείνουμε αυτό το τμήμα της ακρόαση. Δεν έχω το δυνατότητα να δώσω άλλες δυνατότητες λόγου. Πρέπει να περάσουμε στο δεύτερο τμήμα. Δύο-τρία συμπεράσματα μόνο θα συνάξω από τους, τις εμπειρογνωμονές μας. Πρώτον, μία διαπίστωση. Η ζωή είναι μία πολυδιάστατη εμπειρία. Ως εκ τούτου πρέπει να λάβουμε υπόψη κάθε πλευρά της ζωής και να βρούμε μία ισορροπία, κάτι που είναι αναγκαίο σεβασμό της ισότητας μεταξύ άντρα και γυναίκα ένα σημείο μια αφετηρία για να έχουμε μια πιο δίκαιη κοινωνία. Προφανώς με την κρίση έχουμε περισσότερες ε, προκλήσεις και χρειαζόμαστε να δώσουμε διαφορετικές απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται. Να έχουμε μια μεγαλύτερη, μια πιο ευέλικτη αντιμετώπιση της κατανομής των ρόλων ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα. Περισσότερες δημόσιες επενδύσεις για να γίνει πραγματικότητα η ισότητα. Η πολιτική και η κουλτούρα του κόσμου της αγοράς της εργασίας είναι κάτι που πρέπει πάντα να λάβουμε υπόψη μας. Θέλω να κλείσω ευχαριστώντας όσους ε, συνέβαλαν στην συζήτηση και πρότειναν πρωτοβουλίε για το μέλλον. Θα δώσω τώρα τον λόγο και την Προεδρία στη συνάδελφο κύριε Παπαδοπούλου για το δεύτερο κομμάτι της ακρόασης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο χρόνος κυλάει, γι' αυτό θα δώσω το λόγο τώρα στις επόμενες δύο ομιλήτριες του δεύτερου πάνελ και ο τίτλος ε, είναι ε, «Ο συνδυασμός επαγγελματικής και μη επαγγελματικής ζωής». Έχουμε εδώ δύο εμπειρογνωμόνες, την κυρία Ιζαμπέλ Βουέλπε και την κυρία Ανά Ρουμπίν. Να πω λίγα λόγια για τις προσκεκλημένες ομιλήτριες. Η κυρία Ιζαμπέλ Βέλπε είναι πρόεδρος ε, ε, για, στο τμήμα στρατηγικής και οργάνωσης ε, του Τεχνικού Πανεπιστημίου ε, του Μονάχου και έχει σπουδάσει διαχείριση επιχειρήσεων και στην Βοστόνη και στο Πανεπιστήμιο του Μίνστερ και επίσης έχει σπουδάσει στο London School of Economics προτού κάνει το διδακτορικό της, προτού αναλάβει την την έδρα για τη στρατηγική και την οργάνωση εργάστηκε στο ε, Ινστιτούτο Max Planck. Έχει ασχοληθεί με τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και έχει διδάξει ε, στο Πανεπιστήμιο Κλερμόντ, στην ε, Λιόν, το Πανεπιστήμιο Λούτζικ Μαξιμίλιαν και στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης στην Ελβετία. Επίσης, ε, συνεργάζεται με διάφορα επιστημονικά περιοδικά, έχει γράψει αρκετά βιβλία και πολλά άρθρα. Οι έρευνές της ε, έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά. Κυρία Ιζαπέλ Βέλπε, έχετε το λόγο. Δέκα λεπτά έχετε. Δυστυχώ ε, πρέπει να μείνουμε στο χρονοδιάγραμμα. Δύο μιλήτρε έχουμε και θέλουμε να έχουμε και χρόνο για τι ερωτήσει. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Είμαι καθηγήτρια ε, διδάσκω management και θέλω να σας πω πώς οι παγκόσμιες τάσεις ε, θα επηρεάσουν τον τρόπο εργασίας μας και πώς αυτό επιτρέπει καλύτερο συνδυασμό του επαγγελματικού και μη επαγγελματικού βίου. Επίσης ε, μου ζητήθηκε να αναφερθώ σε ε, διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα στο θέμα αυτό. Προφανώς αντιμετωπίζουμε μια σειρά παγκοσμίων τάσεων αυτή τη στιγμή που επηρεάζουν τον τρόπο που οργανώνουμε τη δουλειά μας. Κάτι που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη δυνατότητα συνδυασμού ε, του επαγγελματικού και μη επαγγελματικού βίου. Η πιο σημαντική τάση είναι η παγκοσμιοποίηση. Ποτέ δεν ήταν τόσο διασυνδεδεμένο ο κόσμος. Ε, η πίεση για καινοτομία είναι μεγαλύτερη από ποτέ και βλέπουμε ότι αλλάζουν οι αξίες στον δυτικό κόσμο. Ε, έτσι τώρα λοιπόν δίδεται περισσότερη αξία στην, στον ελεύθερο χρόνο, στην οικογενειακή ζωή. Όλα αυτά ε, σημαίνουν περισσότερη πίεση για τις διάφορες για τις επιχειρήσεις, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να παραμείνουν ε, ε, ανταγωνιστικές. Ταυτόχρονα, χρειάζονται όμως πολύ περισσότερη ευελιξία, πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν σε διάφορες αγορές σε όλο τον κόσμο, πρέπει ε, να μπορούν να αντράξουν τις ευκαιρίες καινοτομία πρέπει να είναι ευέλικτες. Αυτό ζητούν και οι, και εργαζόμενοι. Αυτό σημαίνει ότι ε, το flex security, η ελαστασφάλεια, ευελιξία και ασφάλεια ταυτόχρονα ε, θα πρέπει να παρέχεται και το καλό είναι ότι η νέα γενιά το εκτιμάει αυτό περισσότερο, το να έχει και ασφάλεια και ευελιξία το να μπορεί να συνδυάσει τα διάφορα της δικαιώματα ταυτόχρονα. Από την πλευρά του management, λοιπόν, από την πλευρά της οργάνωσης, ε, βλέπουμε σημαντική καινοτομία στο πώς οργανώνουμε τη δουλειά μας και φυσικά βλέπουμε σε μεγάλο βαθμό τεχνολογική ε, καινοτομία, κυρίως στον τομέα των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής, αλλά βλέπουμε καινοτομία και στον τρόπο που οργανώνουμε τη δουλειά μας ε, και εντός μιας επιχείρησης ε, και οριζόντια. Θα γίνει λοιπόν παράγοντας ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων το θέμα του συνδυασμού επαγγελματικού και μη επαγγελματικού βίου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το επιχειρηματικό μοντέλο ήταν που ε, αποφάσιζε την ε, ανταγωνιστικότητα, ενώ στο μέλλον θα είναι ακριβώς αυτός ο παράγοντας. Ε, η νέα εργασία λοιπόν, να την ονομάσουμε έτσι, τι μορφή θα έχει. Να κοιτάξουμε τις έρευνες που έχουν γίνει. Καταρχάς, προσβλέπουμε στην δημοκρατικοποίηση των επιχειρήσεων. Τον 18ο αιώνα η δημοκρατία ξεκίνησε στον πολιτικό χώρο και αν ρωτούσατε κάποτε, αν, ρωτούσατε τότε κάποιον αν υπήρχε εναλλακτική λύση στη μοναρχία θα σας λέγανε όχι. Είχαν γίνει κάποια πειράματα στη Γαλλία ε, σε κάποιες βρετανικές απικίες ε, στις Πολιτείες αλλά τον 18ο αιώνα ήταν αδύνατο να φανταστεί κανείς ότι θα υπήρχε δημοκρατική εναλλακτική λύση. Παρόμοια ε, ε, επανάσταση, λένε οι προβλέψεις, ε, θα, δούμε σήμερα στις επιχειρήσεις και το βλέπουμε ήδη σε κάποιες επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι ψηφίζουν τη διοίκηση, τη διεύθυνση και αυτό λειτουργεί πολύ καλά. Βλέπουμε ότι πολλές επιχειρήσεις με δημοκρατική δομή, όπως ε, ε, δομή συνεταιριστική, λειτουργούν πολύ καλά. Είναι πολύ ανταγωνιστικές και βλέπουμε ότι απαιτείται πολύ περισσότερη ε, δημοκρατικοποίηση στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον τομέα των ε, επικοινωνιών και πληροφορικής. Αυτή λοιπόν είναι πολύ σημαντική τάση, το ότι οι επιχειρήσεις πια είναι μικρές δημοκρατίες. Έτσι εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες ε, των εργαζομένων σχετικά με το πού θέλουν να εργαστούν, για ποιον και πάνω σε ποια προγράμματα. Η άλλη τάση που βλέπουμε είναι ότι οι επιχειρήσεις ε, πρέπει να ανταποκρίνονται στο, στην απέτηση να είναι σταθερές αλλά και ευέλικτες ταυτόχρονα. Και κάποιες ε, επιχειρήσεις ε, που έχουν πρωτοστατήσει στην καινοτομία είπαν ότι αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο δημιουργώντας μια νέα τάξη εργαζομένων που είναι ελεύθεροι μόνιμοι. Πέρα λοιπόν από τους μόνιμους υπαλλήλους μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει και ανθρώπους ε, από μία ομάδα οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια σειρά προγραμμάτων που μπορεί να προσφέρει η επιχείρηση. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Μπορεί κανείς ε, να το κατακρίνει αυτό θεωρώντας ότι αυτό είναι το τέλος ε, της μόνιμης και ασφαλούς εργασιακή σχέση. Μπορεί όμως κανείς να το θεωρήσει και θετικό, διότι επιτρέπει στον κόσμο να συνδυάζει το ιδιωτικό και επαγγελματικό βίο με πολύ καλύτερο τρόπο, διότι μπορούν να κατευθύνουν πολύ περισσότερο αν θέλουν να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα, αν θέλουν ενδεχομένω ε, να κάνουν ένα διάλειμμα. Ε, μπορούν να έχουν ένα μοσαϊκό απασχόλησης ώστε να αποφασίσουν πόσο χρόνο θέλουν να αφιερώνουν στη δουλειά τους, σε εραστεχνικές δραστηριότητες, στην οικογένειά τους. Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις ε, να μπορούν να πάρουν μια ανάσα και να παρέχουν ε, ευελιξία. Αυτή λοιπόν είναι πολύ σημαντική τάση. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό όσον αφορά τον ε, συνδυασμό επαγγελματικού και μη επαγγελματικού βίου. Η καινοτομία και τεχνολογία μας επιτρέπει να συνδυάσουμε τα πλεονεκτήματα των μεγάλων επιχειρήσεων, ε, για παράδειγμα την οικονομία κλίμακας ε, και πολλά άλλα πράγματα, με τα πλεονεκτήματα μικρών επιχειρήσεων που ξέρουμε ότι η νέα γενιά εκτίμα θέλουν ε, ευελιξία, θέλουν ένα γνώριμο περιβάλλον, λιγότερη ιεραρχία, απασχόληση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μόνο, περισσότερη δημιουργικότητα, καλύτερα κίνητρα. Αυτά παραδοσιακά τα βρίσκαμε σε πιο μικρές επιχειρήσεις. Οι προβλέψεις όμως λένε ότι η τεχνολογία θα επιτρέψει σε όλες τις επιχειρήσεις να συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα των μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. Αυτέ ε, λοιπόν ήταν ε, οι θέσει μου σχετικά με το πώς οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να συνδυάσουν καλύτερα όλα αυτά τα στοιχεία και θα ισχύουν και για άντρε και για γυναίκες. Θα περάσω τώρα στις διαφορές που βλέπουμε. Αποφάσισα λοιπόν να σας δείξω ένα διάγραμμα. Βλέπουμε την κατηγορία διαφόρων επαγγελμάτων όταν σκεφτόμαστε εμείς τα διάφορα επαγγέλματα και τους ανθρώπους, σκεφτόμαστε ωραία πόσο ικανοί είναι οι άνθρωποι αυτοί και πόσο ευγενικοί είναι, πόσο ανθρώπινοι, πόσο μα αρέσουν σαν άνθρωποι. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο διαστάσεις. Όταν ε, λοιπόν γνωρίζουμε κάποιον, ε, συνήθως τον τοποθετούμε κάπου σε αυτόν τον τομέα. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα ένα διάγραμμα για τους άντρες, για τους ανδρικούς ρόλους. Βλέπετε λοιπόν ότι το να είναι κανείς ε, καθηγητής είναι πολύ καλή επιλογή ε, για το επάγγελμά του, διότι βλέπετε ότι είναι πάνω δεξιά, θεωρείται λοιπόν και πολύ ικανός και πολύ ανθρώπινος κανείς. Ζεστός άνθρωπος αυτό είναι καλό, διότι έτσι θα βρει κανείς ε, εύκολα δουλειά και από την άλλη θα θεωρηθεί ότι είναι ότι είναι και καλός άνθρωπος. Στις γυναίκες πώ έχει η κατάσταση. Βλέπετε ότι πάνω δεξιά ε, η περιοχή είναι άδεια. Αυτή είναι η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι άντρε και οι γυναίκες σήμερα όσον αφορά τη συμφιλίωση του επαγγελματικού και του ε, ιδιωτικού βίου. Ε, γιατί, διότι οι γυναίκες που κάνουν σταδιοδρομία ή θα θεωρηθούν ικανές ε, επειδή κάνουν σταδιοδρομία, αλλά όχι ε, ανθρώπινες. Ή θα θεωρηθούν πολύ ζεστοί οι άνθρωποι, αλλά όχι ικανοί. Για να έχει λοιπόν ε, κανείς επιτυχή σταδιοδρομία θα πρέπει να θεωρηθεί ότι τα καταφέρνει καλά και στι δύο αυτέ διαστάσει. Ειλικρινά σα λέω ότι μόλις ολοκλήρωσα ένα μεγάλο πρόγραμμα ερευνητικό πάνω στο θέμα αυτό και το θέμα αυτό δεν είναι θέμα έλλειψης γνώσεων. Συχνά στις έρευνες στην επιστήμη δεν έχουμε αρκετέ γνώσεις. Μπορεί να μην γνωρίζουμε ποιο εμβόλιο είναι καλό κατά μιας ε, ασθένειας, αλλά ε, σε αυτό ε, το πρόγραμμα γνωρίζουμε πολύ καλά όλα τα στοιχεία. Γνωστές είναι και οι λύσεις. Έχουμε όλες τις γνώσεις που χρειαζόμαστε. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί σε μένα, θα του δώσω ε, όλα τα στοιχεία που χρειάζεται. Είναι λοιπόν ε, θέμα εφαρμογής. Ε, είναι μια έκκληση για πολιτικά και θεσμικά μέτρα. Να σας δείξω τα πιο συναρπαστικά αποτελέσματα. Για να συμμετάσχει κανείς σε ένα επάγγελμα πρέπει να υποβάλει αίτηση και ξέρουμε ότι το ίδιο βιογραφικό με, τις ίδιες, ε, με τα ίδια προσόντα ε, αξιολογείται διαφορετικά ανάλογα με το αν είναι βιογραφικό άντρα ή γυναίκας. Κατά τις διαπραγματεύσεις για τον μισθό, οι γυναίκες διαπραγματεύονται μισθό κατά 7% χαμηλότερο και αυτή η διαφορά αυξάνεται. Οι γυναίκες θα πρέπει... Όταν μια γυναίκα επιμένει να πληρωθεί ε, τα ίδια με έναν άντρα τελικά θεωρείται επιθετική και δεν παίρνει τη δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν είναι πιο έξυπνο από πλευρά μια γυναίκα να μην διαπραγματευτεί ε, τόσο σκληρά. Και επίσης το πρόβλημα εδώ πέρα είναι τα στερεότυπα, είναι οι προσδοκίες ε, από τους διάφορους φιλετικούς ρόλους. Αυτό λοιπόν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μέσω διαρθρωτικών μέτρων. Οι καταρτήσεις ε, δεν βοηθάνε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, επί 30 χρόνια προσπαθούν να ασχοληθούν με θέματα ρατσισμού, αλλά το μόνο που βοηθάει στις περιπτώσεις αυτές είναι τα διαρθρωτικά μέτρα. Ε, να συνοψίσω. Η ψηφιοποίηση θα μας επιτρέψει να ε, συνδυάσουμε ε, τα διάφορα μοντέλα εργασίας. Οι εργαζόμενοι θέλουν flex security, θα αυξηθεί δηλαδή η ευελιξία. Αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες που θα δούμε. Θα δούμε επίσης πιο δημοκρατικές και διαφανείς επιχειρήσεις και μπορεί να δούμε και νέα εργασιακά πρότυπα, τα οποία θα πρέπει να στηρίζονται από πρότυπα κοινωνικής προστασίας. Ε, μπορεί δηλαδή να χρειάζονται στήριξη οι άνθρωποι και οι διαφορές ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες ε, συνεχίζουν να υπάρχουν και ξέρουμε ότι οι διαφορετικές, ε, τα ίδια προσόντα αξιολογούνται διαφορετικά ανάλογα με το αν κάποιος είναι άντρας ή γυναίκα. Μόνο διαρθρωτικά μέτρα λοιπόν ε, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν ε, να ε, εξαλείψουν αυτές τις διαφορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Η κυρία Ναρούμπιν, μέλος του Προεδρείου του Ιστερού Κόμματος της Σουηδίας, έχει ασχοληθεί για τη μείωση του χρόνου τα τελευταία χρόνια σπουδάζει νομική, ιδίως δε εργατικό δίκαιο και μόνη της ασχολείται με, την, ε, με τα δικαιώματα των εργαζομένων, των εργαζομένων γυναικών. Ήταν επικεφαλής μια ομάδας εργασίας ε, του κόμματος, του αριστερού κόμματος της Σουηδίας για να εξετάσει το πώς μπορεί να μοιραστεί σε εξάωρες βάδιες η δουλειά στη Σουηδία χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Έχει, πολλές, έχει μιλήσει σε πολλές συναντήσεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και σε συνδικαλιστικές δομές. Είναι μέρος του κόμματος ε, δούλεψε ως συνδικαλίστρια και είναι δασκάλα παρουσίαση των θέσεων των γυναικών σε δημοτικά σχολεία. Την καλωσορίζω και τη δίνω το λόγο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι τώρα. Θα μιλήσω σου ειδιστή. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την ε, Μόλιν Πιόρκ ε, που με κάλεσε. Θα ήθελα όμως ε, να ευχαριστήσω και τις εξαιρετικές ομιλήτριες που άκουσα σήμερα. Η φεμινιστική καρδιά μου νιώθει πολύ καλά όταν ακούω τέτοια πράγματα. Εδώ συζητάμε τα θέματα ισότητας. Δεν θα πρέπει λοιπόν να παραπονιόμαστε για, το, για τους απόντες, αλλά να χαιρόμαστε για τους παρόντες. Εγώ ε, θέλω διατήρηση του μισθού αλλά ε, ε, λιγότερες ώρες εργασίας. Στην γωνία κάθεται ο γιος μου, ο Εμίλιος, ο οποίος με έκανε να σκεφτώ ότι η αξία είναι κάτι παραπάνω από τη δουλειά. Ταυτόχρονα, όταν έμεινα έγκυος, συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι πια ε, τόσο κέρδοφόρα όσο ένας άντρας στην ίδια ηλικία. Και θα μιλήσω για την εργασία. Ξέρουμε ότι η εργασία είναι σημαντική για την ε, διαβίωση, για την κοινωνία, για την ε, παραγωγή προϊόντων, για την ευημερία. Αλλά στον χρόνο εργασίας συμπεριλαμβάνονται και πολλές άλλες έννοιες. Ο χρόνος εργασίας συνδέεται και με την μη πληρωμένη εργασία, με το χρόνο που ε, περνάμε με τις οικογένειές μας ή με το χρόνο που δεν περνάμε με τις οικογένειές μας. Έχουμε το χρόνο που γυμναζόμαστε, που συμμετέχουν σε τέτοιες ε, συνεδριάσεις όπως η σημερινή, ε, τις ώρες που κοιμόμαστε, τις ώρες που κάνουμε, τον κόπο, που κάνουμε τη ζωή να αξίζει. Βλέπετε εδώ πέρα μια ε, παλιά ε, εικόνα ενός ρολογιού, το βλέπετε από το στυλ, αλλά μας ε, δείχνει τον τον διαχωρισμό του χρόνου. Στην Σουηδία δεν εργαζόμαστε 6 ώρες, εργαζόμαστε 8 ώρες. Πολλοί εργάζονται 8 ώρες, άλλοι όμως δεν εργάζονται καθόλου. Υπάρχει λοιπόν ανισορροπία στην αγορά εργασίας. Στην Γαλλία αντιθέτως έχει εισαχθεί μια πιο σύντομη εργασιακή εβδομάδα που διαρκεί 35, εβδομα... 35 ε, ώρες. Και ο λόγος γι' αυτό ήταν να υπάρξουν περισσότερες θέσεις εργασίας και να έχει ο κόσμος ισορροπία ανάμεσα στον ελεύθερο χρόνο και τον επαγγελματικό βίο. Είδαμε ότι οι εργαζόμενοι είδανε βελτίωση του ε, τρόπου διαβίωσης τους ε, και επίσης υπήρχε καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην πληρωμένη και μη πληρωμένη ε, εργασία. Οι άντρε ανέλαβαν περισσότερες ευθύνες στη φροντίδα των παιδιών από την νωρίτερα όταν εργάζονταν 40 ώρες την εβδομάδα, ενώ έτσι περιγράφηκε στι γυναίκες να έχουν άλλες ασχολίες. συνδυασμός ε, της οικογενειακής ε, και της εργασιακής ζωής. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ στα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να λύσουμε το πρόβλημα, διότι εάν ε, δεν υπάρχει νομοθεσία, τότε οι οικογένειες επιλέγουν την παραδοσιακή συνταγή. Οι γυναίκες μένουν σπίτι, είναι πιο ευέλικτες, ενώ οι άντρες ε, ε, θα εργάζονται. Μόλις ολοκλήρωσα μια πανεπιστημιακή εργασία όπου χρησιμοποίησα αυτές τις διάφορες προοπτικές σε δύο συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις. Η μία στόχο έχει την ε, μείωση του χρόνου εργασίας με διατήρηση του ιδίου μισθού, ενώ ε, η άλλη πρόταση είναι να μοιράσουν οι άντρε και οι γυναίκες μεταξύ τους τι μέρες, ώστε οι μητέρες και οι πατέρες να μην μπορούν να ε, δώσουν το δικό τους μερίδιο στον άλλον. Έτσι έχουμε καλύτερη ισορροπία, διότι γνωρίζουμε ότι η εργοδότες πάντα ε, θα κάνουν διακρίσεις εις βάρος των γυναικών όσο αυτές μένουν σπίτι κατά παράδοση για να ασχοληθούν με τα παιδιά ε, και όσο εκείνες συνήθως ε, έχουν θέσεις μερικής απασχόλησης. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να λύσουμε το θέμα στη βάση τους ώστε οι εργοδότες να μην έχουν πια κίνητρο για να κάνουν διακρίσεις. Εδώ βλέπετε στοιχεία από τη Σουηδία. Βλέπουμε ότι μερική απασχόληση έχουν κατά 32% οι γυναίκες ε, στη Σουηδία, ενώ ε, το 10% μόνο των ανδρών. Επίσης βλέπουμε ότι 77% των γυναικών ε, παίρνουν γονεακή άδεια, ενώ το 23% των ανδρών, παρότι η σουηδική νομοθεσία προβλέπει ίσο μοίρασμα. Και εδώ βλέπετε τον ε, φαύλο κύκλο ανισοτήτων. Οι γυναίκες εργάζονται με μερική επασχόληση, έτσι έχουν ε, χαμηλότερη αμοιβή. Γι' αυτό δεν μπορούν να πάρουν διαζύγιο, διότι εξαρτώνται οικονομικά, παρότι μπορεί να μην είναι ευτυχισμένε. σε κάτι που οδηγεί ε, στο να αναλάβουν την βασική ευθύνη για τον οικοκυριό, το οποίο σημαίνει ακριβώς ότι δεν μπορούν να πάρουν μια θέση ολικής απασχόλησης, πλήρους απασχόλησης. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ισότητα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εργαζόμαστε 6 ώρες την ημέρα με τον ίδιο μισθό. Το συμπέρασμα μου είναι ότι η μείωση του χρόνου εργασίας ε, αυτή καθ' αυτή δεν θα οδηγήσει σε ισότητα. Η ε, οι σκληρότεροι επικριτέ λένε ότι οι άντρε, αν έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο, θα πάνε να πίνουν μπύρε ή να βλέπουν ποδόσφαιρο. Μπορεί αυτό να είναι αλήθεια, αλλά. Και έτσι, μάλιστα, οι γυναίκε θα πρέπει να λάβουν ακόμα περισσότερο την ευθύνη για τα παιδιά ή για το νοικοκύριο. Γνωρίζω ότι οι προτάσεις μου ε, ε, είναι επίμαχες, ε, αλλά αν μοιράσουμε το χρόνο εργασίας ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες και μειώσουμε το χρόνο εργασίας, τότε δημιουργούνται ίσες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση της της οικογενειακής ζωής. Καταλαβαίνω ότι σε 10 λεπτά είναι δύσκολο να τα πει κανείς όλα. Φαντάζομαι ότι θα θέσετε ερωτήσεις μετά. Πολύ ευχαρίστω θα σας στείλω τις εργασίες που έχω εκπονήσει. Εδώ βλέπετε μία, δύο φωτογραφίες. Η πρώτη προέρχεται από το 1973, όταν στη Σουηδία καταργήθηκε η εργασία το Σάββατο. Από 48 ώρες την εβδομάδα ε, περάσαμε σε 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Βλέπετε λοιπόν ε, μία οικογένεια που κάνει πικνίκ, πίνει καφέ Σάββατο πρωί, επειδή δεν χρειάζονται πια να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Το 2020 έχουμε πέμπτη απόγευμα που η οικογένεια πηγαίνει για πικνίκ στο πάρκο. Επειδή εργάζονται μόνο έξι ώρες την ημέρα. Αυτό λοιπόν είναι το όραμά μας. Αφού το καταφέραμε στο παρελθόν μπορούμε να το ξανακαταφέρουμε. Και θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την ε, σουηδική πολιτική και ποιο είναι το νόημα της πολιτικής. Ο Ούλοφ Πάλμε, ε, Σουηδός Πρωθυπουργός, δολοφονήθηκε, αλλά τα λόγια του παραμένουν, παρότι ε, ήμουνα μόλις έξι ετών όταν πέθανε. Η πολιτική δεν έχει μόνο να κάνει με, τον προϋπολογισμό, έχει να κάνει με τη βελτίωση της ε, ζωής των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να τολμήσουμε να έχουμε ένα όραμα για την εργασιακή ζωή όπου να υπάρχει ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είμαι πολιτικός, γι' αυτό θα αναφερθώ στην κατάσταση σήμερα, ε, θα αναφερθώ στην, στην ε, σημερινή κυβέρνηση στη Σουηδία. Ε, βλέπουμε ότι μειώνει τη φορολόγηση για τους πλούσιους, ενώ ενώ υπονομεύονται τα δικαιώματα και οι παροχές για τους πιο φτωχούς. Ποιε θα είναι λοιπόν οι οικονομικέ συνέπειε μια ημέρα εργασία που να κρατάει 6 ώρε. Μερικοί πιστεύουν ότι θα επανέλθουμε στην εποχή του λίθου και δεν θα έχουμε πια ανάπτυξη. Αλλά η έκθεσή μας δείχνει ότι με αν είχαμε μόνο τις μισές περικοπές ε, φόρων που έχει εφαρμόσει σήμερα η κυβέρνηση, θα μπορούσαμε να έχουμε ε, αυτή την ε, ημέρα σε έξι ωρών. Η πολιτική λοιπόν έχει να κάνει με την πολιτική βούληση. Αυτό λοιπόν ήταν το συμπέρασμά μου. Τρία δευτερόλεπτα βλέπω ότι μου μένουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και μια καλή συζήτηση. Ευχαριστώ. I thank you very much as well. Ευχαριστώ και για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Λίγοι ευρωβουλευτέ είναι πλέον παρόντε και δεν υπάρχουν ερωτήσει. αλλά αν κάποιο θέλει το λόγο, μπορεί να θέσει ερωτήσει. Να πείτε ποιοι είστε. Και κάντε ερωτήσεις παρακαλώ, γιατί μόνο 10 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας συνολικά. από την Επιτροπή Γυναικών της ε, Ένωσης Συνδεδομικών της Εύρωσης, το Μετρό του Λονδίνου. Είπετε ότι όταν μείνετε έγκυος γίνεται λιγότερο παραγωγική, αλλά εγώ πιστεύω ότι γίνεσαι περισσότερο γιατί παράγεις ένα νέο άνθρωπο. Και το θέμα του προβλήματος της ισορροπίας είναι ότι η ισορροπία της αποδόπλευρας δεν έχει οικονομική αποτίμηση, αλλά δεν είναι έτσι. Η οικογενειακή ζωή είναι δουλειά, δουλειά αγάπης, αλλά δουλειά που πρέπει να αναγνωρίζετε Η ισορροπία λοιπόν καλό είναι, αλλά καλύτερα είναι να πούμε για συλλογικοποίηση της δουλειάς αυτής. Γι' αυτό γίνεται μέσω βρεφονιπιακών σταθμών, ε, κοινωνικής πρόνοιας, εθνικών υπηρεσιών που προστατεύουν αυτές τις δομές. Αυτές είναι που περικόπτουν οι κυβερνήσεις με τα προγράμματα λιδωτότητας. Και οι γυναίκες είναι αυτές που πληρώνουν το τίμημα της μείωσης του κόστους αυτού. Αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη. Μετά για την Ιζαμπέλ. Είπατε ότι οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι θέλουν flexicurity. Αλλά μήπως άλλο πράγμα εννοεί ο ένας άλλο ο άλλος. Οι εργαζόμενοι θέλουν μια ασφαλή θέση εργασίας και φέτος και του χρόνου να σέβεται ο μισθός το κόστος, ε, ε το κόστος ε, εργασίας. Αλλά οι εργοδότες θέλουν να εκμεταλλεύονται όσο περισσότερο γίνεται για όσο περισσότερες ε, ώρες μπορούν τους εργαζόμενους με όσο λιγότερο μισθό γίνεται. Γι' αυτό βλέπεις ε, αύξηση άτυπων ε, συμβάσεων εργασίας που διευρύνουν το, και, τις αποκλήσεις ε, μισθών λόγω φύλου και το ότι οι γυναίκες μπαίνουν σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος? Να πείτε ποια είστε. Πίτερσεν λέγομαι. Από την... Ε, το Γερμανικό Συνδικάτο συνδικαλιστών. Έχω μία ερώτηση. Γίνονται γίνεται έρευνα για τον ανταγωνισμό που μπορεί να προκύψει μεταξύ εργαζομένων. Οι γυναίκες δεν θα μπορούσαν να μετάσχουν σε ένα έργο στο μόναχο για την κινητικότητα. Έχει γίνει κάποια τέτοια σχετική μελέτη. Άλλη μια ερώτηση, αν θέλετε. Παρακαλώ. Από την H Platform Europe. Πρώτος άντρας είμαι που παίρνει το λόγο. Βλέπω με χαρά ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνδρες εδώ. Ευχαριστώ όλους όσοι υπογράμμισαν τη σημασία της ε, μέρημνας και τη σύνδεσή τους με τις συντάξεις. Ο φορέας μου προστατεύει τα δικαιώματα των ηλικιωμένων και βλέπουμε ότι στην πολύ μεγάλη ηλικία ιδίω οι ηλικιωμένε γυναίκες δεν είναι σε καλή κατάσταση. Έχουν μικρές συντάξει διότι ήδη από το ξεκίνημα ήταν μικρότερες καθότι πολλές, η δουλειά που κάνουν στην κοινωνία συχνά δεν πληρώνεται ούτε υπολογίζεται στο ΑΕΠ ή στα συστήματα εισφορών όταν πεθάνει ο άντρας τους μπορεί να μην έχουν δικαιώματα πολλά ή κεφάλαιο για να αντιμετωπίσουν τα τελευταία και πιο ακριβά χρόνια της ζωής τους. Αναγνωρίστε, θα ήθελα να αναγνωρίσετε το ζήτημα των συντάξεων και της ανάγκης να υπολογιστεί ο τρόπος προστασίας των παιδιών και των ηλικιωμένων. Παρακαλώ τις δύο, τα δύο μέλη του πάνελ να απαντήσουν. Ε, Just be brief because we have only a few minutes. Okay. Yes. Και να είστε σύντομες. Θα συνεχίσω στα σουηδικά. Ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα. Είναι η γλώσσα που μιλάω καλύτερα. Ε, να ξεκινήσω από την κυρία από τη συνδικαλιστική οργάνωση. Δεν έπιασα το όνομά σα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ με όλα όσα είπατε. Καλά, τώρα μιλάω αγγλικά, αλλά δεν πειράζει. Ναι, όχι, συμφωνώ με όλα όσα είπατε. Και εγώ όταν ήμουν 24 ετών ε, ε, ε, ήμουνα στην ίδια κατάσταση. Δεν ήθελα να είμαι ευέλικτη, ήθελα να έχω σταθερή θέση εργασία. Δεν ε, με ενδιέφερε να αλλάξω χώρα, να ανταγωνίζομαι με άλλους εργαζομένους. Ήθελα ασφάλεια, όχι ευελιξία. Είναι λοιπόν λίγο μύθος το ότι, ο κόσμος, ότι οι νέοι θέλουν να είναι μόνο ευέλικτοι. Επίσης, όσον αφορά τις γενικές συλλογικέ λύσεις, και ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να παρέχουν την απαραίτητη προστασία. Όσον αφορά λοιπόν την ανταγωνιστικότητα και το ότι οι γυναίκες δεν μπορούν τελικά να είναι τόσο ε, ευέλικτες, ε, συμφωνώ ότι ε, το flexicurity αποτελεί κίνδυνο για τις γυναίκες. Είναι λοιπόν πολύ καλό το ότι το συζητάμε και προς τον τελευταίο κύριο που αναφέρθηκε στην φροντίδα των ηλικιωμένων. Χαίρομαι που το αναφέρετε, διότι δεν πρόλαβα να το πω αυτό στην ομιλία μου. Όταν οι γυναίκες εργάζονται με μερική απασχόληση και φροντίζουν ε, ε, τους ε, συγγενείς τους στο σπίτι τους, αυτό δεν επηρεάζει μόνο το μισθό, επηρεάζει και τη σύνταξή τους. Με την πρότασή μας για εξάωρο την ημέρα, οι γυναίκες που σήμερα εργάζονται με μερική απασχόληση, σημαίνει ότι αυτό πια θα θεωρείται πλήρης απασχόληση και έτσι θα αυξηθεί και ο μισθός τους. Είναι λοιπόν ε, πολύ σημαντική αυτή η πρόταση. Ε, φοβάμαι ότι δεν έχω χρόνο να απαντήσω σε άλλες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Yes. θα μιλήσω στα σουηδικά, αν ε, μου επιτρέπετε, διότι ήταν δύσκολες οι ερωτήσεις όσον αφορά το flexicurity, την ελαστασφάλεια. Γνωρίζουμε ότι Ε, κάποιες επιχειρήσεις ε, δεν μπορούν να βρουν εξειδικευμένο προσωπικό. Απ' την άλλη υπάρχει η διορθωτική ανεργία. Αυτό το μοντέλο λοιπόν δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλο για όλες τις επιχειρήσεις ε, και για όλους τους τομείς. Αλλά οι επιχειρήσεις βλέπουμε ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ευέλικτα πρότυπα. Η ε, ανησυχία σας είναι ότι αυτό θα οδηγήσει σε εκμετάλλευση. Η ε, τεχνολογία επικοινωνίας και πληροφορική όμως ε, επιτρέπει διαφάνεια στο βαθμό που δεν είχαμε ποτέ. Έτσι λοιπόν ε, μπορούμε να ελέγξουμε πώς φέρονται οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους. Μπορεί να στιγματιστούν οι κακοί εργοδότες σε το employer branding και έτσι να μην βρίσκουν πια εργαζομένους. Επίσης, στις νέες αυτές μορφές που θα χρησιμοποιούνται από το μέλλον, που ζητούν οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να υποστηριχθούν ε, από νέα πολιτικά μέτρα, για παράδειγμα ένα βασικό εισόδημα, ώστε να παρέχεται αυτό που ζητάνε και οι επιχειρήσεις ε, και οι εργαζόμενοι. Ε, να υπάρχει δηλαδή ασφάλεια, αλλά και μόνο ασφάλεια δεν κάνει ευτυχισμένο τους ανθρώπους. Το 70% των εργαζομένων δεν είναι ικανοποιημένοι στην ε, δουλειά τους. Ε, θέλουν ε, περισσότερη ευελιξία, περισσότερη ομαδική εργασία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αυτό πώς μπορεί να εφαρμοστεί από πλευρά της διοίκησης των επιχειρήσεων. όσον αφορά τις έρευνες, πρόκειται για νέα μοντέλα. η ΖΕΜΚΟ, η έχουν καταργήσει την διεύθυνση και οι εργαζόμενοι μόνοι τους οργανώνονται και εγώ ως επιστήμον θεωρώ ότι θα είναι αντικείμενο ερευνών το να δούμε αν θα έχουν επιτυχία. Είναι σχετικά νέα αυτή η εξέλιξη και γι' αυτό σας την ανέφερα σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. I think here we can uh, Ευχαριστώ. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτό το πάνελ και θα μιλήσω ελληνικά τώρα. Ζούμε σε μια εποχή κρίσης και οπωσδήποτε αυτή η κρίση έχει και πολλές κοινωνικές προεκτάσεις στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών περιμένουν πολλά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περιμένουμε και εμείς οι γυναίκες αρκετές πολιτικές που θα αντιμετωπίσουν ακριβώς τα πολλά δημοκρατικά ελλείμματα, τα στερεότυπα, τις ανισότητες. Σήμερα μιλήσαμε για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Αν δούμε το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης ή του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα συρτάρια υπάρχουν πάρα πολλά directives, υπάρχουν οδηγίες, υπάρχουν νομοθεσίες. Η ουσία είναι μια. Με τα μέτρα λιτότητα τα οποία σήμερα λαμβάνονται και πλήττουν ανεπανόρθωτα των κοινωνικών ιστών, κυρίως στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, στην Πορτογαλία από όπου προέρχεται η συνάδελφός μου η Ρετζίνα Μπάστος, στην Κύπρο από όπου προέρχομαι εγώ, στην Ελλάδα από που προέρχεται μια άλλη ομιλήτρια, η κυρία Δανάκη εάν λάβουμε υπόψη ότι αυτά τα μέτρα λιτότητος αυτή τη στιγμή κατασπαράσουν ουσιαστικά ό,τι έχουμε πετύχει ως Ευρωπαϊκή Ένωση και χτυμένα εργατικά και κυρίως στο θέμα της ισότητας των φύλων ουσιαστικά φαίνουν ένα πισωγύρισμα γιατί όταν υπάρχει ανεργία, όταν υπάρχει φτώχεια, όταν υπάρχει ε, αλυσιδωτές και υπάρχει έξαρση της βίας στην ίδια την οικογένεια οι απειλέ είναι εδώ και μεγάλη, το μεγάλο στίχημα που έχει η ευρώπη αυτή τη στιγμή εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών των ευρωεκλογών του μαΐου του 2014 είναι ότι βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. παίζει μεγάλο ρόλο ποιοι θα εκλεγούν για ευρωβουλευτέ, τον Μάιο και ποιοι θα είναι αυτοί οι νέοι ηγέτε οι οποίοι πραγματικά θα προωθήσουν τι πολιτικέ λιτότητα και θα δουν πώ να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα τη θηλυκοποίηση τη φτώχεια, τη θηλυκοποίηση τη ανεργία, τη θηλυκοποίηση τη βία, τη θηλυκοποίηση όλων αυτών των κοινωνικών αρνητικών επιπτώσεων που έχουν τα αρνητικά μέτρα λιτότητα και δυστυχώ και πολλέ φορέ οι άδικε αποφάσει που λαμβάνουν λαμβάνονται στο eurogroup πίσω από κλειστέ πόρτε. γιατί η τρόικα αγαπητοί φίλοι και φίλε δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση δεν λογοδοτεί σε εθνικά κοινοβούλια δεν λογοδοτεί στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. επομένω καταλήγοντα είμαι ευτυχή γιατί προέδρευα σε αυτό το πάνελ ευχαριστώ όλου του πολύ εκλεκτού ομιλητέ που ήταν όλε γυναίκε ευχαριστώ και του άντρε του ακροατηρίου που είχαν την υπομονή να βρίσκονται εδώ και κάποιοι να πούν και τι δικέ του ερωτήσει ο δρόμος για την ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς είναι μακρύς αλλά το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο είναι εδώ γιατί είναι ο μόνος θεσμός της ευρώπης που εκλέγονται οι ευρωβουλευτές από τα εκατομμύρια των λαών της ευρώπης τα 500 εκατομμύρια πολίτες και ως εισηγήτρια του ευρωπαϊκού έτους πολιτών που ήταν το 2013 χαιρετίζω ακριβώς την πρόταση της επιτροπής φαμ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου το 2014 να είναι έτος συμφιλίωσης οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων γιατί μόνο αν όλοι μαζί δουλέψουμε ώστε να αυξήσουμε το awareness το ενδιαφέρον των πολιτών και αν δουλέψουμε να έχουμε ενεργούς πολίτες που στέκουν κριτικά και ζητούν να συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε τότε μπορούμε να ελπίζουμε. και θα καταλήξω σε κάτι. έχω ακούσει την ομιλήτρια να μιλά σε αυτό που έχει πει ο ο νέος Σουηδός Πρωθυπουργός για το θέμα τη βελτίωση των πολιτών, ότι χρειάζονται να γίνουν πολλά. Εγώ θα πάω πολλέ πολλούς αιώνες πριν όταν οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι που είχαν βάλει και τη βάση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας είχαν μπει και ειδικά ο Σοκράτης να επιδιώκει στη βελτίωση της ζωής των πολιτών αυτή ήταν η φράση του Σοκράτη. Γιατί είναι αδύνατο να βελτιωθεί ο κόσμος αν δεν βελτιωθεί πρώτα ο άνθρωπος. Ζούμε μια οικονομική κρίση. Η κρίση αυτή δεν είναι μόνο ε, πώς να ευημερήσουν οι αριθμοί και οι άνθρωποι να παίρνονται. Ζούμε μια κρίση που πρέπει να την ταυτίσουμε με μια κρίση αξιών. Και αν θέλουμε να πάει μπροστά η κοινωνία θα πρέπει να ξεκινήσουμε ακριβώς πώς να βελτιωθεί πρώτα ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος σημαίνει άντρα και γυναίκα. Πώς οι πολιτικέ συμφιλίωσεις, η βελτίωση της ζωής των γυναικών να είναι το στίχημα που πρέπει να κερδίσει η Ευρώπη και αυτό είναι το μεγάλο στίχημα που πρέπει να να κερδίσουμε κι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις επόμενες εκλογές αναδεικνύοντας άντρες και γυναίκες ευρωβουλευτές που πράγματι θα είναι αγωνιστές για αυτά τα θέματα ισότητας. Εδώ κλείνω. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τις ομιλήτριες που ήταν όλες εξαιρετικές τη συνάδελφο μου κυρία Ρετζίνα Μπάστος. Εύχομαι στους βουλευτίνες και στους βουλευτές που θα τρέξουν για τις επόμενες ευρωεκλογέ να καταφέρουν να κερδίσουν και να συνεχίσουμε από αυτά τα έβρονα, όλοι μαζί ξανά, εύχομαι το ειδόν και για μένα, αυτήν την πάλη για την ισότητα των φύλων. Και το στίχημα είναι να καταφέρουμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη, γιατί είναι πολύ σημαντικό, οι περικοπές που γίνονται λόγω των πιέσεων που δέχονται να μην είναι στον τομέα της υγείας και της παιδείας διότι η υγεία και η παιδεία είναι δύο νευραλγικοί τομείς που αν πραγματικά μειώσει τα κονδύλια σημαίνει ότι δεν έχουμε προοπτική για μια καλύτερη και βαθύτερη Ευρώπη. Και αυτή είναι η δική μας επιδίωξη γιατί αγαπούμε την Ευρώπη και θέλουμε την Ευρώπη να αντέξει σε αυτές τις πιέσεις και να γίνει ε, να γίνει πιο κοντά στον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια σε όλους. Ε, ευχαριστώ πολύ και όλους τους ε, διερμηνείς και επίσης τη γραμματεία των δύο επιτροπών ε, και Employment που στήριξαν όλη αυτή τη συζήτηση σήμερα. Ευχαριστώ θερμά. Muito brevemente, também umas últimas palavras para Και εδώ να κλείσω την συνάντηση και εγώ από πλευρά με δύο λόγια. Μια πολύ χρήσιμη συνάντηση. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο για να έχουμε μια καλύτερη, ένα καλύτερο συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Η συζήτηση δημιουργεί δύο προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Την δημογραφική, το δημογραφικό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί και το πρόβλημα της οικονομικής ανάπτυξης. Η μεγαλύτερο ή μικρότερο πρόβλημα, ιδίως στις χώρες ε, που αντιμετωπίζουν κρίση. Χρειάζονται λοιπόν πολιτικά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίπεδο κρατών μελών για να αντιμετωπίσουμε τις δύο αυτές προκλήσεις στις πολιτικές που πρέπει να διαμορφώνονται με σωστό τρόπο κάθε μέρα. Έχουμε μια μεγάλη ευθύνη σήμερα και στο μέλλον. Η πρόκληση είναι να εξασφαλίσουμε ισότητα μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών για να έχουμε μια πιο δίκαιη κοινωνία. Μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες που ζητούν οι πολίτες από τους πολιτικούς και αυτό διαπιστώθηκε με συγκεκριμένη μελέτη που έγινε πρόσφατα είναι να καλυφθεί το, ε, το μισθολογικό χάσμα και να καλυφθεί και όταν θέλουμε να καλύψουμε με καλύτερο τρόπο, την να ισορροπήσουμε με καλύτερο τρόπο οικογένεια και δουλειά, μπαίνει και το θέμα του μισθολογικού χάσματος στο παιχνίδι. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τι ζητείτε να κάνουμε για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Σωστά αναφέρθηκε από πολλές εμπειρογνώμονες ότι πρέπει να απαντούμε σε παγκόσμιες προκλήσεις και στις κοινωνικές αλλαγές που βλέπουμε και που απαιτούν μια διαφορετική οπτική από την μερική απασχόληση, την προσωρινή απασχόληση, την ε, κατανομή των ευθυνών σε οικογενειακό επίπεδο. Ας αδράξουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή. Πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις τέθηκαν. Ευχαριστώ και καλό απόγευμα.